Οπότε έχουμε την έκθεση Τάνοκ. Κύριε Τάνοκ, έχετε να πείτε κάτι ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα είπα χθες το βράδυ, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Το βασικό πρόβλημα τις τελευταίες μέρες με τις συμβαστικές τροπολογίες και καταφέραμε να διαπραγματευτούμε αρκετές ήταν η συμβαστική υπαρτιμών 13 για το ζήτημα του ότι σημειώνουμε το αίτημα της Σομαλιλάνδης να ζητήσει αναγνώριση ως κράτος. Το σημειώνω μόνο χωρίς να το κρίνω, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες για τη διαδικασία, γιατί το ΕΛΚ από ό,τι φαίνεται δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και από ό,τι κατάλαβα συζητώντας με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής θα συζητήσουμε επί της ε, τροπολογίας αυτής και μετά θα υπάρξει μια ξεχωριστή τροπολογία επί της ε, τροπολογίας της για να διαγραφεί οποιοδήποτε αναφορά της Ομαλιλάνδης. Αυτό είναι ατυχές το ότι μπορούμε να σβήσουμε μία από τις μεγάλες προκλήσεις ε, εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή για το ζήτημα της Ομαλιλάνδης. Δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή, Κανένα δεν ασχολείται σοβαρά με το ζήτημα χωρί να αναφέρει αυτό το θέμα και ειλικρινά απευθύνω έκκληση στο ΕΛΚ ε, να αναθεωρήσει την στάση του. Ε, όπως το έχω διατυπώσει είναι τελείως ουδέτερο και η διάσκεψη του Λονδίνου που ήταν η βασική διάσκεψη για τη Σομαλία νωρίτερα φέτο, ανέφερε ρητό στο ζήτημα τη Σομαλιλάνδη και πρέπει το ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα μεταξύ Μογκαντήσου και Χεγγέισα και δεν είναι δυνατόν να το σβήνουμε εντελώς. Αυτά τα δήλωσαν ηγέτες από όλο τον κόσμο και νομίζω πως η θέση του ΕΛΚ εδώ πέρα δεν είναι λογική. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 75 υπέρ, κατά Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Την τροπολογία 75. Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Αν ψηφίσουν ε, ΕΛΚ και σοσιαλιστές και όλας. Λοιπόν, πέρας. Έγινε δεκτή λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 77 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 79 σε δύο μέρη. Μέχρι το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές δεκτών. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90, 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ συμβαστική 105 μάλιστα 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και περνάμε. Τι έχουμε εδώ, κάτι καινούριο. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής 6α. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 123 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές Δεκτεί. 123 μέρος δεύτερο υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 7 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 129 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 130. Να επαληθεύσουμε. 129 δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Γίνεται δεκτή. 38 με 10. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην τροπολογία 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 131 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 132 υπέρ κατά αποχές αυτή. Η σοσιαλιστική ομάδα αν ψήφιζε έτσι κάπως πιο τακτικά θα ήταν καλό. Μα δεν ψηφίζεται όλη η ομάδα, δεν ψηφίζει. 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 136 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 142 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 144 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 147 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 148 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 154 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 156 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 168 υπέρ κατά αποχές δεκτή 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 100 όχι συμβαστική 13 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Ωραία. Check then. Compromesso 13. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 176 υπέρ 176 Καλώς, περνάμε τότε στην 179. 179 εβδομήντα εννέα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκατόν εβδομήντα εννέα. Πέρας της φοφορίας 31 με 15 και μία εποχή γίνεται δεκτή λοιπόν 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 187 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 198 υπέρ. 189 με συγχωρείτε, κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 191 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε στη 205 υπέρ κατά αποχές δεκτή 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή 211 υπέρ κατά αποχές δεκτή 214 υπέρ κατά αποχές δεκτή 215 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 28 Η 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 30 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 31 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ, το πρώτο μέρο, κατά αποχές δεκτή, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 38 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 39 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 40 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 48 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 49 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 50 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 51 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 52 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 53 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή μπορούμε από 63 μέχρι 71 να τις ψηφίσουμε μαζί από 63 μέχρι 71 υπέρ. Κατά. Καλώς. 63 μέχρι 69 πλήν 68 υπέρ. Μα είπε ότι θέλει χωριστή ψηφοφορία στο 69. Μέχρι το 79 λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. 69 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή από την 3 μέχρι τη 12 μπορούμε να τη ψηφίσουμε μαζί γιατί όχι. 2 υπέρ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά légge αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά Δέβε 5 ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Der Antrag ist 28. Εγκρίνεται λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική, άρχιτη ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Και η έκρηση, η έκρηση εγκρίνεται με 42 ψήφους υπέρ, 6 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν. Charles, περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η κυρία Γιαννάκου είναι η Μαριέτα, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι. Περνάμε άρα συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ένα υπέρ κατά ορίστε στην 8 οπότε πέρας της ψηφοφορίας ναι Περνάμε στην τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια για να... Ε, Μαριέτα. Περνάμε τώρα στην έκθεση πρόοδου για το Μαυροβούνιο. Schon wieder hat der Kollege Tenok das Wort. Και πάλι τον λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ. Ich bitte doch die Kollegen auf den billigen Plätzen ruhig zu sein. Εκεί πίσω στα ορεινά στις τινές θέσεις κάντε λίγο ησυχία. Mr. David, I understand you, but... <laughs> David, σας καταλαβαίνω, αλλά... So, Charles, du hast das Wort. Mr. Tenok, the floor is yours. Κύριε Τάνοκ, έχετε το λόγο. Hmm? Mr. Tenok, would you like to start? Θα θέλω, κύριε Τάνοκ. Ψυχία παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Right, Mr. Chairman. Μάλιστα, λέει ο κύριος Τάνοκ. Μαυροβούνια, Πρόεδρε. Υποψήφια χώρα από το Δεκέμβριο του 2010. Και τώρα έχουν αρχίσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις βαλκανική χώρα ε, προχωρεί, προοδεύει όσον αφορά, και, ε, όσον αφορά την ένταξη. Το μικρό είναι όμορφο, πολλές φορές λέμε, αλλά εδώ πέρα είναι μπερδεμένη η χώρα ε, και πάντοτε δεν έχουμε ξεκάθαρη διάκριση εξουσιών. Έχουμε θέματα οικογενειών που κυβερνούν τη χώρα, αλλά τέλο πάντων υπάρχει γενικά συνένεση ε, από τι πολιτικέ δυνάμει για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω χωρίσει σε πέντε τμήματα την έκθεσή μου. Πρώτα-πρώτα έχω τι γενικέ εκτιμήσει που λέμε ότι εκφράζουμε ικανοποίηση για τι ε, εκλογέ ελεύθερε και ειρηνικέ πολιτικά κριτήρια μετά και είπαμε ότι υπάρχει τώρα το δικαίωμα ε, στο κεφάλαιο 23 όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ασφάλεια ε, τα κεφάλαια αυτά ε, θα είναι προκλήσεις για τη χώρα, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Σουηδία που θα υποβάλουν βέτο για την αρχή των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την ε, προσχώρηση. Πάντως είναι σοβαρή τουλάχιστον στις δηλώσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, αλλά βέβαια στα Δυτικά Βαλκάνια αυτό το πρόβλημα είναι πάγιο και ενδυμικό. Ε, μετά έχουν πολιτικά κριτήρια, λέμε ότι χρειάζεται να κατοχυρωθεί ανεξαρτησία δικαστικής αρχής, τον, ε, η, κοινωνία των πολιτών, ε, τα τα Ε, όλα αυτά θα πρέπει να αναβαθμιστούν και είχαμε όσον αφορά πηλές προς δημοσιογράφους για ε, εκεί πέρα ένα θέμα. Επίσης υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη μεταχείριση των μειονοτήτων ε, εθνοτικές μειονότητες, ε, επιθέσεις εναντίον ε, λεσβιών, ομοφυλοφίλων κλπ. Και Επίσης υπήρχε κάποιος πολιτικός, ο οποίος υπέστη πάρα πολύ καταπίεση, η μία ήταν ομοφιλόφιλος. Ε, επίσης ε, από το 2011 έχει αρχίσει η πορεία της χώρας προς ε, τον ΠΟΕ και θα πρέπει να δούμε το ότι χρειάζεται να ασχοληθούν στη χώρα αυτή με περισσότερους τομείς της οικονομίας πέραν του τουρισμού. Να μεταρρυθμιστεί η αγορά της εργασίας. Εξαρτάται από το ευρώ η χώρα παρά το ότι βέβαια το Μαυροβούνιο δεν ανήκει στην Ευρωζώνη, αλλά χρησιμοποιεί τον ευρώ σαν σημείο αναφοράς και όπως είναι σήμερα η κατάσταση αυτό είναι προβληματικό. Πάντως το τι είναι αδύνατο το ευρώ βοηθά τον τουρισμό στη χώρα. Και βέβαια δείχνουν πρόθυμοι να νομοθετήσουν ε, εκεί που χρειάζεται, αλλά βέβαια το θέμα είναι και να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Συνεργασία, διμερείς, διμερείς ζητήματα υπάρχουν, έχει καλή σχέση η χώρα με τους ε, γείτονε. Είναι πρωτοπόρο το Μαυροβούνιο όσον αφορά ε, την περιφερειακή συνεργασία και ιδίως με την Κροατία γίνεται μετάφραση του κοινωνικού κεκτημένου. Σε σχέση με τη Σλοβενία επίσης προχωρούν οι επαφές της χώρας. Και βέβαια βοηθά το ότι υπάρχει κοινή γλώσσα ε, μεταξύ των χωρών ή της οικογένειας των δημοκρατιών της πρώην ε, Γιουγκοσλαβίας. Πέρσι Είχαμε συνθήκε με Σερβία, Μακεδονία, Κροατία που συνήψε η χώρα και αυτό διασκέδασε κάποιες ε, ανησυχίε που υπήρχαν για τους εγκληματίες, τους Σέρβους που είχαν ε, καταφύγει και είχαν κρυφτεί στο Μαυροβούνιο. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει αυτοί οι εγκληματίες, οι Σέρβοι, να μην κάνουν πια ε, αυτό το πράγμα, να μην προσφεύγουν στη χώρα του στο Μαυροβούνιο. Και κατοχυρώθηκε το ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Παραπέμφθηκαν κάποιοι για διαφθορά και επίσης υπάρχει και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, μια υπόθεση, αλλά καλά πάνε τα πράγματα στη χώρα και κάποιοι μυρογνώμονες θεωρούν ότι εκτός από την ε, Κροατία οι υπόλοιπε χώρες Δυτικών Βαλκανίων θα αργήσουν να ενταχθούν. Έτσι όπως είναι σήμερα η πολιτική συγκυρία. Να δούμε βέβαια τι θα προβλέπει η νέα συνθήκη για το 2016 και μετά. Εν πάση περιπτώσει κάνουν αυτά που χρειάζεται οι Μαυροβούνιοι και εγώ δεν μπορώ παρά να θεωρήσω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη χώρα στην ευρωπαϊκή διαδρομή της. Κούκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να καλωσορίσω την έκθεση του κύριου Τάνοκ. Είναι πάρα πολύ συνεπές, συνεπής και έχει περιλάβει σχεδόν όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν το Μαυροβούνιο. Πολύ σημαντική βάση και καλή βάση για τη συζήτηση. Θα ήθελα σύντομα να αναφέρω κάποια θέματα που αναφέρονται και στην έκθεση. Πιστεύω πως είναι σωστά εστιασμένη η έκθεση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τις εσωτερικές υποθέσεις, το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά καθώς και θέματα που σχετίζονται με την δημόσια διοίκηση και την οικοδόμηση δυνατοτήτων για διαπραγματεύσεις. Η εστίαση σε αυτό το τομέα θα είναι πολύ σημαντική για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερα χρειάζεται η ενίσχυση της, του δικαστικού ε, σώματος για την καταπολέμηση κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ε, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η δίωξη των ε, υποθέσεων διαφθοράς. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να ενισχύσει τις διοικητικές και ε, Ε, κοινωνικές του δομές. Επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε επαφέ με την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τα θέματα του, της ένταξης, τα πρωταξιακά. Ε, ε, νομίζω πως από ό,τι κατάλαβα μάλλον η κοινωνία των πολιτών έχει εκπροσωπηθεί στις διαπραγματεύσεις και συμμετέχει άμεσα στις ε, διαπραγματεύσεις αυτές. Ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να μιμηθούν και οι υπόλοιπε χώρες. Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τους Μαυροβούνιους για την εξαίρετη διεξαγωγή των εκλογών. Η νέα κυβέρνηση έχει μια φρέσκη και ισχυρή εντολή για να δουλέψει πάνω στην ατζέντα της ε, Ένωσης και θα πρέπει να επενεθεί για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Eh, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ καταρχήν Να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνο για το τελευταίο κείμενο που μας παρουσίασε. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση λοιπόν αναφέρει ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από πλευρά Μαυροβουνίου. Υπάρχει, υπάρχει λοιπόν πρόοδο, χαιρετίζουμε τι ελεύθερε και δημοκρατικέ εκλογέ και διαπιστώνουμε πως έχει ενισχυθεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Και εδώ πέρα λοιπόν πρόοδος. Και επίσης ε, τα προβλήματα στα ΜΜΕ. Αυτός ήταν ε, ένας τομέας στον οποίο είχαμε ασκήσει κριτική στην τελευταία έκθεση και εδώ πέρα έχουμε πρόοδο. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς ε, και επίσης πρέπει να αναλυθούν κάποια μέτρα για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προωθηθεί η συμμεταχείριση. Δεν έχω να προσθέσω άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Θα υποβάλω λοιπόν κάποιες τροπολογίες και νομίζω πως και άλλες ομάδες θα κάνουν το ίδιο. Και χαίρομαι που με τον Τσάρλς. Η κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και μάλλον να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την έκθεσή του. Δίνει μια πολύ ακριβή και περιεκτική έκθεση για την κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Είμαι επίσης ευτυχής που έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία σε αυτό το σώμα που στηρίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας διεύρυνσης στο Μαυροβούνιο και θα έχουμε μία επαφή με, αύριο με βουλευτές σε μια διακοινοβουλευτική δηλαδή επιτροπή ε, και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να δούμε και πάλι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του κυρίου Τάνο. Και εγώ θέλω να σχολιάσω δύο σημεία το ένα είναι ότι ίσως θα ήταν καλό να αναφέρουμε το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο στο Σύνταγμα του αναφέρεται στον εαυτό του ως μια οικολογική χώρα. Πράγμα που στην πράξη δεν είναι αλήθεια σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα για τα μεγάλα projects στον τουρισμό αλλά και στην παραγωγή ενέργειας πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδος εδώ αλλά το να αναφέρεστε σε κάτι που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα μπορεί να στηρίξει τους Μαυροβούνιους όντως να γίνουν πιο οικολογική χώρα. Και όλοι συμφωνούμε για το γεγονός ότι η Κομισιόν θα ξεκινήσει 23-24 ε, Δεκεμβρίου το πρόγραμμα, ιδιαίτερα γιατί για την διαφθορά υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν στο δικαστικό κλάδο, και στην κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα της διαφθοράς και αυτό είναι σημαντικό για τη διαδικασία. Είμαι ευτυχής που ο κύριο Τάνοκ ήδη έχει περιλάβει τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Έγινε μια ακρόαση την περασμένη εβδομάδα νομίζω, όχι πριν δύο εβδομάδες για τη διαφάνεια στη διαδικασία διεύρυνσης και εκεί δόθηκαν κάποια αρκετά καλά παραδείγματα που ανέφεραν διάφοροι Κροάτες για το πώς τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα στο μέλλον. Και άρα λοιπόν ίσως θα ήταν καλό να συμπεριληφθούν και κάποια παραδείγματα για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Για τον ε, ρόλο εποπτείας του, του Κοινοβουλίου ε, ξεπλάγει ευχάριστα την περασμένη εβδομάδα όταν είχαμε μια επαφή με τον πρέσβη του Μαυροβουνίου όταν προετοιμάζαμε την ε, αυρινή συνεδρίαση. Τρεις πρόεδροι των τριών ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν προκύψει από κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το Κοινοβούλιο το ίδιο. Κύριε Τάνοκ, τώρα εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στο θέματα των LGBT, των ομοφιλόφιλων και άλλων. Και θα ήθελα να αναφερθεί στην έκθεση το γεγονός ότι η ίδια κυβέρνηση, παρότι υπάρχει πολύς ε, φόβος απέναντι στους ομοφυλόφιλους στη χώρα, έχει φτιάξει ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης και έχει κάνει και μια περιφερειακή διάσκεψη για τα θέματα των νομοφιλόφιλων την άνοιξη φέτος. Υπάρχουν όντως προβλήματα στη χώρα, ε, συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση και την κοινότητα των νομοφιλόφιλων και τον, την κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα θέματα τα οποία προωθούν. Εν γέννη όμως είναι πολύ καλή έκθεση και θα μπορέσουμε πολύ ωραία να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να συμφωνήσω με όλα τα θετικά που είπαν οι προλαλήσαντες και να σχολιάσω επίσης αυτή τη σύντομη αλλά ουσιαστική έκθεση του κυρίου Τάνοκ. Νομίζω πως ένα από τα χαρακτηριστικά της κατάστασης στο Μαυροβούνιο, που είναι πολύ θετικό, είναι ότι έχει επιτευχθεί ευρεία διεθνή συνένεση όσον αφορά την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα πολιτικά κόμματα. Και δεύτερον χαρακτηριστικό είναι ότι η κοινωνία των πολιτών πολύ επιτυχώς ενεπλάκει στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και φαίνεται πως το Μαυροβούνιο επιτυχώς θα ανοίξει και θα κλείσει κάποια κεφάλαια όταν θα, θα φτάσουμε στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Επίσης θα ήθελα να τονίσω πως τα θέματα διαφθοράς που είναι βέβαια σημαντικά αλλά και αλλού, όχι μόνο εκεί, ε, έχουν μειωθεί σημαντικά γιατί η κοινωνία ανησυχεί Και έχουν, έχουν γίνει μάλλον πολύ συγκεκριμένα βήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα με τις γειτονικέ χώρες, που δεν είναι όμως πολύ σοβαρά και αντιμετωπίζονται εν μέρη. Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά θέματα στις διμερείς σχέσεις, ειδικά ο η χάραξη των συνόρων είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το φροντίσουμε προσεχώς, γιατί διαφορετικά θα προκύψει πρόβλημα. Να πω επίσης ότι το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο τα καταφέρνει από μόνο του να προσεγγίσει την Ένωση να πω όμως ότι το μέλλον και η μοίρα του εξαρτάται και από τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν, ο συντονισμό και επαφέ ανάμεσα σε όλε αυτέ τι χώρε και τι κυβερνήσει τη περιοχή χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρουσα η έκθεση που μας ε, κατέθεσε ο κύριος συνάδελφος, πιο προσεκτική θα έλεγα και πιο αντικειμενική στην παρουσίαση των γεγονότων. Ε, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα που ίσως να μην είναι της έκθεσης, άλλα τα περιλαμβάνει, άλλα δεν τα περιλαμβάνει. Είναι προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και μας για την πραγματική εικόνα που παρουσιάζει αυτό το μικρό κράτος των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και για την προσπάθεια που πρέπει να γίνει να αντιμετωπιστεί το πρώτο θέμα και σωστά επικεντρώνουμε την προσοχή μας είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο. Όμως ε, έχω την εντύπωση αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν είναι η κλασική βαλκανική διαφθορά μόνο, λαθρεμπόριο λοιπά γνωστές υποθέσεις, επειδή η χώρα ακολουθεί μια πολιτική, θα έλεγε κανείς, ιδιωτικοποίησεων και ξεπουλήματος, θα έλεγα εγώ, του φυσικού πλούτου, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων στο ξένο κεφάλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εμπειρία μου λέει ότι έχουμε ή μπορούν να παρατηρηθούν φαινόμενα διαφθοράς. Επομένως υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα. Αυτές οι εταιρείε αυτοί που έχουν εξαγοράσει αυτά τα, το φυσικό χώρο, την τουριστική ανάπτυξη, οι υπηρεσίες, τι φόρο αποδίδουν στο κράτος του Μαυροβονίου, ώστε να έχει κάποια ωφέλη και αν αυτά τα, η φορολογία ε, μεταφέρεται σε κοινωνική πολιτική, εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό ερώτημα διότι δεν είναι μόνο η πλευρά που έθιξε η συνάδελφος από τους πράσινους ότι θα μπορούσε να ήταν πιο περιβαλλοντικό. Θα έλεγα ε, η προσπάθεια των κυβερνήσεων για μετατροπή σε τουριστικό παράδεισο ε, φοβάμαι ότι το έχει ε, πάει να το μετατρέψει σε ένα χώρο εύκολης κερδοφορίας των ξένων επενδύσεων και επιδείνωση της ε, κατάστασης στην κοινωνία του Μαυροβουνίου. Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα, νομίζω δεν αναφέρεται η έκθεση, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το ποσοστό της ανεργίας των ε, εργαζομένων στο Μαυροβούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που είδα, έχει αυξηθεί, αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά και έχει φτάσει περίπου 12,98-13%. Είναι υψηλό ποσοστό. Φυσικά στις εποχές που ζούμε έχουμε ευρωπαϊκές χώρες νυν μέλη με υψηλότερα ποσοστά, αλλά δεν είναι καλό σημάδι. Και επομένως υπάρχει ένα θέμα τι γίνεται και ποιες πολιτικές ακολουθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστεί, επαναλαμβάνω, το θέμα της ανεργίας και το θέμα της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων ηλικιών, χαρακτηριστικό που συνοδεύει τη μεγάλη ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Τρίτη παρατήρηση, θα ήθελα να αναφέρεται η έκθεση, θα κάνουμε σχετικές τροπολογίες, και σε προβλήματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δημόσια αγαθά, η έμφαση που θα με ενδιέφερε και θα μας ενδιέφερε και ενδεχομένως καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες είναι τα θέματα της παιδείας, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Παρατηρείται, ενδεχομένως να μην συμβαίνει στην ίδια έκταση, ότι το πρόβλημα αυτό, αν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, ιδιαίτερα τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, και αναφέρομαι γιατί κουβεντιάζουμε, έχω την έκθεση της Αλβανίας, είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Επομένως η έκθεσή μας, ε, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, εγώ νομίζω πως είναι έτσι, πρέπει να δώσει έμφαση και σε αυτά τα θέματα, γιατί πραγματικά μια ενταξιακή διαδικασία που σημαίνει πίεση εντατικές προσπάθειες πρέπει να έχει και ωφέλη για το λαό και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Ε, θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε με τον κατάλογο των σκιωδών με τον συνάδελφο Χούντι. Έχω ακόμα δύο συναδέλφους μόνο. Τον κύριο Πέτερλε, και σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε την Κίνα και το Ιράκ και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Άρα, πρώτο ο κύριος Πέτερλε και μετά ο κύριος Κατσίν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω το λόγο. Λόγω της κοινή μας ιστορίας με το Μαυροβούνιο. Αλλά θέλω να έχουμε κοινό μέλλον. Όντω έχουν πετύχει πρόοδο σε διάφορου τομεί. Παρ' όλα αυτά όμω θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο όσον αφορά το κράτο δικαίου, όσον αφορά την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο ε, να καταφέρουν να έχουν λιγότερη διαφθορά και να βελτιωθεί και η διοίκηση. Ο Κάτσιν. Κύριε Πρόεδρε, το Μαυροβούνιο είναι η μικρότερη χώρα της ε, περιφερειάς μας. Ήταν βέβαια και στην πρώην Ιουγκοσλαβία η μικρότερη δημοκρατία. Σήμερα πάντως θεωρείται πρωτοπόρος χώρα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων μετά την Κροατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια άλλη τέτοια φιλόδοξη χώρα η οποία θέλει ε, να έχει ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Ήδη έχει ανοίξει δύο κεφάλαια η χώρα αυτή ε, και προ του τέλους του έτους θα έχει ανοίξει και το κεφάλαιο 25 σε σχέση με έρευνα και επιστήμη. Νομίζω ότι όπως άνοιξε νωρίς θα κλείσει και νωρίς. Θα πρέπει να δούμε καλά ότι στην περιοχή έχει σταθεροποιητικό ρόλο η χώρα αυτή. Θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι θα συμβάλλουν στην σταθερότητα της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, που είναι πολύ σοβαρό, πρόκειται να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Σερβίας και τον πρόεδρο του Κοσμοπεδίου, την κυρία Γιάεβα δηλαδή και τον κύριο Νίκολης. Ποτέ σε τέτοιο επίπεδο δεν είχε γίνει διάλογος. Πριν από λίγα χρόνια αποσχίστηκε τον Ρουμούνια από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Είναι σημαντικό όλο που έχουν διαδραματίσει, πρέπει να του συγχαρούμε γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να συγχαρούμε σίγουρα και τον εισηγητή. Είναι υψηλή ποιότητα η έκθεσή του και ελπίζουμε ότι ε, αυτή τη βδομάδα που θα συναντήσουμε την προσωπία του Μαυροβουνίου θα έρθει και ο κύριο Τάνακα μαζί. Κύριε Λάγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε που με καλέσατε και που με αφήνετε να σχολιάσω ε, τα της έκθεσης ε, νομίζω ότι ε, η έκθεση λέει ότι λέει και η δική μας έκθεση πρόοδο. Αυτή που δόθηκε στη δημοσίευση τον Οκτώβριο. Νομίζω επίσης ότι δίνουμε ένα μήνυμα έτσι. Έχουμε πει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση της χώρας να εστιάζεται εστιάσει την προσοχή της στα θέματα της ε, ατζέντα ένταξης, να συνεχιστεί ε, αυτή η κομματική συνένεση όσον αφορά τα σημαντικότερα ε, σημεία που αφορούν την ένταξη. Και βέβαια έγιναν εκλογές, έχουμε, θα έχουμε τώρα μια, ένα, μια καινούργια κυβέρνηση θα λάβει όπου να είναι τα καθηκοντά της. Κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να κάνουν επίση είναι το να ψηφιστούν οι σχετικές θεμελιώδεις διατάξεις για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αυτό τα λέει και το ψήφισμα, αλλά επίσης θα πρέπει να σας ε, ε, επιβεβαιώσω ότι, ότι έχουμε ικανή εκπροσώπηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών ε, στους φορείς λοιπόν που λαμβάνουν ε, μέρος στην μεταρρύθμιση της χώρας και τελευταίο που να σας αναφέρω αφορά τα διμερεί ζητήματα. Υπάρχει έντονη ενθάρρυνση να επιληθούν τα προβλήματα με τις γειτονιάρουσες χώρες. Αυτό είναι και δική μας πολιτική, θέλουμε να συνεχιστεί η προτεραιότητα που δίνει σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να σας ε, πω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και η, το, το, το screening, η εξέταση των ζητημάτων συνεχίζεται. Θα ολοκληρωθεί τον ε, Ιούνιο του 2013. Επίσης έχουμε ήδη και κάποιες εκθέσεις ε, screening για τα κεφάλαια 23 και 24 που έχουν φτάσει στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου σημειώνεται πρόοδος και η Προεδρία πρόκειται να καλέσει τους Μαυροβουνίους ούτως ώστε να προπαρασκευαστούν τα προγράμματα δράσης για να δρομολογηθούν για το πρώτο ήμιση του 2013. Επίσης έχουμε και πρόοδο στο κεφάλαιο 25 που αφορά την έρευνα και σύντομα θα ζητηθεί στο Συμβούλιο. Εάν δεν υπάρξει αρκετή πρόοδος προς τα τέλη του έτους, τότε πρέπει να έχουμε μια διακυβερνητική διάσκεψη στις 18 Δεκεμβρίου για να διαπιστωθεί το πόσο έχει προοδεύσει η χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Τάνοκ για να κάνει τα τελικά του σχόλια, ήθελα να θυμίσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Τάνοκ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σύντομα. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου που είπαν καλά λόγια για την έκθεση και εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω την γραμματεία που με βοήθησε. Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα αλλά που προχωρά προς σωστή κατεύθυνση. Δέχομαι τα σχόλια της κυρίας ε, Λούνα Τζέκο για το ότι είναι οικολογική χώρα. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πολιτικά πάντοτε ένα δύσκολο παζάρι ανάμεσα σε οικονομικούς πολιτικούς στόχους και οικολογικούς στόχους. Ε, είναι δύσκολη η απόφαση που θα πρέπει να τη λάβει η κυβέρνηση του, Μαυροβουνίου. Για είπε ο τα είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, η Κροατία δεν θα μπει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χωρίς να έχει λυθεί το θέμα των σύνορων. Για τον Έλληνα συνάδελφο, τον κύριο Χουντή, η ανεργία είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα και η στατικική για την ανάπτυξη και η παιδεία είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και όσον αφορά τον ανεξάρτητο, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ε, όλοι ξέρουν όλους εκεί πέρα είναι τόσο μικρή η χώρα που το να πει κανείς πως δεν γνωρίζει τον δικαστή μάλλον θα είναι ψέμα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει απόλυτη αμεροληψία και ακαιρεότητα σε μια τόσο μικρή χώρα. Πάντως δουλεύουν σκληρά κάνουν ειδική κατάρτιση για όλους τους δικαστές. Και όσον αφορά τώρα τα σχόλια του κ. Κατζίνη για τη συνάντηση με τους ε, ε, βουλευτές του Μαυροβουνίου, θα είμαι πίσω την Πέμπτη από το Βερολίνο και θα έχουμε επαφή μαζί τους. Ε, σας ευχαριστώ πάντως για την υποστήριξή σας και πραγματικά πιστεύω πως το Μαυροβούνιο θα πάει μπροστά. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. επόμενο θέμα είναι οι σχέσεις με την Κίνα, τις Ένωση με την Κίνα. Ο κύριος Μπάσιαν Μπέλτερ, ο εισηγητής, είναι παρόν. Να θυμίσω πως η έκθεση της ΑΦΕΤ δεν ασχολείται με τα θέματα που καλύπτονται από την έκθεση της ΙΝΤΑ, Ευρώπη και Κίνα και ισορροπημένο εμπόριο. Η έκθεση που εθετήθηκε από το Κοινοβούλιο 23 Μαΐου, του 2012 αποφάσισε ήταν να μην δώσει γνωμοδότηση για την έκθεσή μας. πάση περιπτώσει, κάποια μέλη έχουν καταθέσει τροπολογίες που σχετίζονται με το εμπόριο. Και δεδομένης της εξαίρεσης των θεμάτων περιεμπορίου από αυτή την έκθεση, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και από την διάσκεψη των Προέδρων, θα πρέπει να ε, ακόμα και αν υποβληθούν για ψηφοφορία θα θεωρηθούν απαράδεκτες οι σχετικές τροπολογίες. Να μειώσουν λοιπόν οι συνάδελφοι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ήδη αναγνωρίσει το θέμα και επέσυραν τις ε, τροπολογίες αυτού του είδους. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και θυμάμαι ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν η 9η Οκτωβρίου το μεσημέρι στις 12. 333 ε, ε, τροπολογίες ελήφθησαν εντός προθεσμίας, εμπρόθεσμα και ο εισηγητής έχει κάνει 21 συμβαστικέ. Δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπέλτερ να μας πει την ε, γνωμοδότησή του. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις 333 ε, τροπολογίες που δείχνουν το ενδιαφέρον σας για το αντικείμενο της έκθεσης, της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Συζητήσαμε καλά με τους κυριώδεις εισηγητές ε, ε, από τις ομάδες και καταλήξαμε σε 21 συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες ε, οι οποίες βασίζονται στα εξής εκτιμώντας και παραγράφους εκτιμώντας α, g, h, i, l, n και o και στις παραγράφους 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 και 18 Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψατε μου να αναφέρω ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, χτες το βράδυ έλαβα ένα email για την ε, συμβαστική τροπολογία 10 όπου η Άλντε έκανε μια πρόταση αλλαγής της και αφορά την ε, CCP θεωρώντας πως έχει κάποια ευρεία λαϊκή αποδοχή. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοεί εδώ πέρα η σκιώδηση ε, Νομίζω ο συντονιστής των σοσιαλιστών ήδη έχει ήδη Κάτι άλλο αφορά τις ειδικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Είναι ένα υποκεφάλαιο που αφορά τις εμπορικέ ε, ε, σχέσεις. Και βέβαια εδώ πέρα συμπεριλαμβάνουμε και συμβαστική τροπολογία. Υπάρχει λοιπόν μια ξεχωριστή παράγραφος για το ιστορικά πολύ ευαίσθητο θέμα αλλά και οικονομικά και εμπορικά πάρα πολύ σημαντικό. Να αναφέρουμε τις εντάσεις ε, αυτό το καλοκαίρι για τις διάφορες εδαφικές ε, διαφορές και έχουμε σε συνεννόηση με τους πιο καταλήξει στην ε, συμβαστική τροπολογία 20. Επίσης υπάρχει μια προφορική τροπολογία Επίσης, ε, γίνεται λόγος για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κίνας ε, εν μιλάμε για το ότι θα πρέπει η κίνηση του ότι έχουμε ανταποκριτές κινέζικων μίμιε στην Ευρώπη να σημαίνει από την άλλη μεριά πως θα έχουμε και Ευρωπαίους ε, ανταποκριτές οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ε, στην ε, Κίνα, στο Πεκίνο και στο Τοντσίν. Είχαμε και συναντήσεις με την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στην Κίνα οι οποίοι μας είπαν πως δυστυχώς το κλίμα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 υπήρχε μια χαλάρωση από πλευράς κοινοζικών αρχών όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των ξένων ανταποκριτών και πέρσι και φέτος, ε, από ό,τι μας είπαν και μας παραπονέθηκαν, η ελευθερία για να συγκεντρώσουν ε, ειδήσει ε, περιορίστηκε σημαντικά και θα ήθελα και εδώ πέρα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία σχετικά. Οπότε ελπίζω να μπορέσετε να την δεχτείτε ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω επίση να τονίσω πως οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και είναι εκτός των συμβαστικών ε, τροπολογιών βεβαίως θα κρυφτούν και θα εμφανιστούν στις ε, λίστες ψηφοφορίων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη μέχρι τώρα συνεργασία και αναμένω την ε, προσοχή σας. Ε, first on my list of speakers, Mr. Ο κύριος Κασουλίδης, σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ. Mr. President, first of all, I would like to... Κασουλίδης, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπέλτερ διότι ετοίμασε μια πάρα πολύ ισορροπημένη έκθεση, ακριβώς όπως ε, θέλει και το Κοινοβούλιο, να εκθέτει τις απόψεις του. Και για την Κίνα και για τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για την συνεργασία του με τους ε, σκιώδεις ηγητές. Κάλυψε τις περισσότερες μας παρατηρήσεις. και επίσης κατέληξε σε 21 συμβαστικές τροπολογίες. Με αυτές εμείς συμφωνούμε. Οφείλω επίση να σας πω ότι σε σχέση με την πρόταση Watson, νομίζω ότι ήταν ο κύριος Watson που έχει υποβάλει αυτή του την πρόταση για την τροπολογία υπαριθμών 10, θα ήθελα να πω ότι και με αυτό το σημείο συμφωνούμε. Επίσης, Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε ούτως ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι, πιο, πιο σταθεροί όσον αφορά κάποιες ε, περιπτώσεις που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και να δούμε τι θα γίνει με την προφορική τροπολογία που αφορά τα ΜΜΕ. Πάντως και επί της αρχής δεν διαφωνούμε. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εμπορικές σχέσεις, για άλλη μια φορά υιοθετήσαμε δίκαιες απόψεις δηλαδή είπαμε ότι θέλουμε ενιαία πολιτική προς την Κίνα και προς ενιαία Κίνα ούτως υπήν αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους πυράβλους τους που απειλούν από πλευράς Κίνα και αυτό δεν, δεν βοηθά αυτές οι απειλητικοί κατά της Ταϊβάν πύραυλοι. Επίσης, θεωρούμε ότι η Ταϊβάν δικαιούται του να έχει ουσιαστική παρουσία στα διεθνή φόρα. Τώρα όσον αφορά την διαμάχη για τις νήσους και εδώ φροντίσαμε να έχουμε ίσες αποστάσεις από τις δύο χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Εξωτερική Υπηρεσία συγκεκριμένα δεν παίρνουν το μέρος κανένας. Πάντω επ' αυτού έχω κάποια επιφύλαξη για αυτήν την νέα παράγραφο που έχει εισαγάγει ο συγητής και εκεί χαιρετίζει την ε, ε, πρωτοβουλία του Προέδρου της Ταϊβάν όσον αφορά την διαμόρφωση μια συνένεσης για κάποιο κώδικα διοντολογίας όσον αφορά την ε, θάλασσα της Κίνας και βέβαια δεν διαφωνώ με το προηγούμενο αλλά θεωρώ ότι με αυτή τη διάταξη ερχόμαστε σε αντίθεση με αυτό το οποίο είπαμε, δηλαδή ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ίσες αποστάσεις από όλους τους εμπλεκομένους για την διαφορά για τις νήσους. Τέλος πάντων, ε, εγώ θα το συζητήσω ε, στην συνεδρίαση της πολιτικής μου ομάδος και την πέμπτη θα σας πω κατά πόσον θα ε, επιψηφίσουμε ή όχι τη σχετική παράγραφο επί της οποίας βάλει την επιφύλαξη. Κατά τα άλλα πάντως νομίζω ότι ήταν πολύ αξιόλογη η οχι τη σχετικη παραγραφο επι της που βαλει την επιφυλαξη κατα τα αλλα παντως νομιζω οτι ηταν πολυ αξιολογη η δουλεια μας και πάρα πολύ αξιόλογα τα αποτελέσματα. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή αξιόλογη έκθεση και με την συνεργασία και με τους ε, σχεδοσυγητές και άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε κυρία Μπέλτερ. Κυρία Κοπά. Thank you, Mr. President. Η σημερινή συζήτηση δείχνει για μία ακόμα φορά την πολυπλοκότητα του ζητήματος και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν ε, στο, στην Επιτροπή, πράγμα που φαίνεται και από το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Ε, είναι σαφές και προκύπτει και σε έρευνες που γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες ότι η Κίνα προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι σχέσεις με την Κίνα είναι σύνθετες και θα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν και μέσα από αυτό το, την έκθεση και μέσα από αυτή την έκθεση καταφέρουμε να εκφραστούμε με μια ενιαία φωνή. Η σχέση που θέλουμε να οικοδομήσουμε με την Κίνα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στα ζητήματα αρχών και αμοιβαία στα ζητήματα εμπορίου. Η σχέση είναι αλληλένδετη, για να μην δημιουργεί όμως ερωτήματα και ανησυχίες, πρέπει να έχουμε το κουράγιο να βάλουμε τα δύσκολα θέματα στο τραπέζι. Επομένως, στη σημερινή πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι σαφές ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για το θέμα των αρχών είναι επίση σαφές ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κίνα είναι σημαντική για την Ευρώπη, ειδικά σήμερα. Όμω θέματα όπω η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο η θρησκευτική ελευθερία, όλα αυτά που αποτελούν τον πυρήνα των αξιών και των αρχών της Ένωσης πρέπει να μπουν επιτακτικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά ζητήματα, πνευματικά δικαιώματα, ε, απομιμήσεις προϊόντων ή φαρμάκων, το dumping, η χρήση απαγορευμένων ε, χημικών ουσιών, αυτά όλα βλάπτουν σοβαρά την ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και απειλούν την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και φυσικά το περιβάλλον. Άρα, για την οικοδόμηση μιας ισότιμης εταιρική σχέσης, η Κίνα οφείλει να ενταχθεί στα διεθνή πρότυπα και να τα σεβαστεί. Και σε αυτό το πνεύμα θα παρακαλούσα τον εισηγητή να καταρτήσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες του. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλτερ για τη συνεργασία και να επικεντρωθώ τώρα σε μία συμβαστική τροπολογία, την οποία αναφέρει και ο ίδιος, δηλαδή την υπαριθμόν 10. Σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία πρέπει να ομολογήσω πως υπάρχει μια θέση που μας είναι πολύ δύσκολη. Στην αρχή της παραγράφου μιλάμε για το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας το οποίο ε, θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως ε, έχει έχει μεγαλύτερη αποδοχή μεταξύ των πολιτών παρά το ότι αυτό δεν έχει επαληθευθεί από ελεύθερες εκλογές. Από πού μπορεί να ξέρει κάτι τέτοιο άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν δεν υπάρχει δημοκρατική επιβεβαίωση. Πώς το επαληθεύσαμε εμείς χωρίς εκλογές. Απόδειξη το ότι αποδέχεται ο Κινέζικος λαός στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ε, δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά αναφέρουμε πως ε, η αποδοχή αυτή από τον Κινέζικο λαό διακινδυνεύει τώρα λόγω της διαφθοράς, της έλλειψης ε, της έλλειψης διαφάνειας και της κόκκινης αριστοκρατίας. Μα ε, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να ανησυχούμε για την αποδοχή του ΚΚ της Κίνας, αλλά είμαι σίγουρος πως οι τρεις λόγοι οι οποίοι αναφέρονται μάλλον δείχνουν έλλειψη αποδοχής η οποία επιβεβαιώνεται εκατομμύρια φορές κάθε μέρα στο ίντερνετ. Και αναρωτιέμαι αν ε, πραγματικά θα πρέπει ε, αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε αυτή την προσεκτική κριτική που αναφέρεται εδώ πέρα, τα μιλάμε για διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας κτλ. Ε, όταν στην αρχή ε, εγκρίνουμε την ε, κατάσταση και εκδίδουμε μια βεβαίωση, εάν θέλετε, η οποία δεν ξέρω από πού προκύπτει και νομιμοποιείται. Ευχαριστώ τον λόγο έχει ο κύριος Τάνο, καλά σα παρακαλέσω να είστε γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα πριν έρθει ο πρέσβης τον είπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπέλτερ για την εξαιρετική του έκθεση σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα τη σχέση με την Κίνα. Πρέπει να δηλώσω κάποια συμφέροντα εδώ πέρα. Είμαι πρόεδρος της ε, ομάδας φιλίας με την Ταϊβάν, οπότε με ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στο στενό της ε, Ταϊβάν μεταξύ της ε, Κινέζικης Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και χαίρομαι για το ότι μιλάτε για ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας. Ε, βεβαίω η Κίνα είναι ένα οικονομικό φαινόμενο ε, και σημαντικό είναι να έχουμε διάλογο με αυτό τον παγκόσμιο οικονομικό γίγαντα αλλά παραμένει μια μονοκομματική κομμουνιστική δικτατορία. Αν και βεβαίω κομμουνιστικό δεν μου φαίνεται το να πληρώνει κανείς υγεία και παιδεία, αλλά τέλος πάντων ε, ναι, μην ξεχνάμε πως είχαμε και την πρόσφατη δολοφονία ενός Βρετανού πολίτη που έλεγε πολλά σε όσους παρακολουθούν ε, τα της Κίνας όπως επίσης και τη μεταβάση της εξουσίας στον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Οπότε εξελίσσεται η Κίνα αλλά το εάν πηγαίνει προς μια φιλελεύθερη κατεύθυνση είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σαφώς ε, εξακολουθούν να υπάρχει υψηλό επίπεδο παραβίασης και απαράδεκτο ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων εκτελέσεις ε, ε, βίες ε, εκτρώσεις, ε, ακόμα και φήμες για συλλογή οργάνων από πιστούς του Φαλούν Γκόγκ, επιβολή όρκου στο πίστη στο Κινέζικο κόμμα στη δικαιοσύνη. Οπότε δεν υπάρχει κάτω δικαίου παρά μόνο πίστη στο Κομμουνιστικό κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε σχέση με την Κίνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως και τις ε, δυνάμεις της, ε, της ασκή στην περιοχή σε συνοριακές διαφορές με το Βιετνάμ, την Ινδονησία, Μπρουνέι, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα κτλ. Οπότε προβληματική η κατάσταση. Αλλά η μεγάλη, μεγάλη μου ανησυχία είναι η στήριξη για τις σκληρές δικτατορίες ε, της Βόρειας Κορέας, Λευκορωσίας, Σουδάν, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τη Ρωσία συντάχθηκαν με τους, για τη Συρία φυσικά συντάχθηκαν με τους Ρώσους. Και φαίνεται πως υπάρχει μια σκλήρινση της ε, γραμμής τους ε, τους ε, τελευταίους μήνες και αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Γιατί βεβαίως κάηκαν στο χειλό με την αποχή από τη Λιβύη και δεν θέλουν να το επαναλάβουν. Όπως είπα λοιπόν τώρα τα οικονομικά τους ε, συμφέροντα επεκτείνονται στην Νότια Αμερική, σε ολόκληρη την Αφρική, μεταλλευτικά. Οπότε στηρίζουμε τις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες ως ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνο και κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. είμαι σύντομη και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπέλτερ για την έκθεσή του αλλά και για την καλή θέληση που έδειξε και η θέληση συνεργασίας ε, με τους συναδελφούς των πολιτικών ομάδων οπότε και καταλήξαμε σε αυτές τις εύστοχες ε, συμβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να σας τονίσω ότι και εμείς ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ε, νέα αντιμετώπιση, νέα γλώσσα για την Ταϊβάν. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι αυτά τα οποία είπαμε για τα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα ε, πέρασαν. Πέρασαν γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις με τη χώρα αυτή. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε το τι γίνεται από τους ε, Κινέζους και τι γίνεται και από τις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Τι κάνουν δηλαδή στην Κίνα, ε, αγωνώντας τελείως τα εργασιακά δικαιώματα, καταπατώντας τα δικαιώματα φυλακισμένων, ανηλίκων κλπ. Επίσης θέλω να σας πω ότι προσωπικά επίσης συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Μπουτικόφερ. το Κοινοβούλιο δεν είναι εις θέση να κρίνει την ανταπόκριση, το, το, το έρισμα τέλο πάντων στην κινέζικη κοινωνία του ΚΚΚ. Και κατά τη γνώμη μου, το πιο σωστό θα ήταν α, αυτό το τμήμα της παραγράφου της Συμβασικής ε, Πρωτοβουλίας να, να, ε, να απαλληφθεί. Και επίσης σε πλευρά της πολιτικής μας ομάδα θα με τον κύριο Μπέλτερ. Ευχαριστούμε κύριε Γκόμες. Όχι, δεν θέλω τώρα να. δεν θέλω εγώ τώρα να επιστρέψω λεπτομέρειε. Απλώ θέλω να σα πω κάτι, ε, ένα θέμα αρχή. Συνήθω, όταν προσπαθούμε να προγραμματίσουμε την πολιτική μα με κάποιον συνομιλητή, με κάποιον σημαντικότερο, όπω είναι η Κίνα, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να καταλάβουμε εμεί τι συμφέροντα έχουμε στι σχέσει αυτέ και επίση το, το τι συμφέροντα έχει και η άλλη πλευρά στι σχέσει μαζί μα. Τώρα, δεν θέλω να επικρίνω τον κύριο Μπέλτερ, πάρα πολύ αξιόλογο έργο επέτελεσε. Αλλά είναι παραδοσιακό μα λάθο το να αγνοούμε το, το, το συμφέρον τη άλλη πλευράς και να προσπαθούμε να, να, να, του, να, του, να του πούμε, να του, να του για το τι πρέπει να αλλάξει στι πολιτικέ που ακολουθεί. Και ε, αν δεν υπάρχει επομένω συνένεση, τελικά καταλήγουμε να τονίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και σωστά και τα θα τα προσέχουμε γιατί είναι οι αξίες μας τις οποίες και πρέπει να προωθούμε όμως ποτέ θα μπορέσουμε τις αξίες μας να τις ε, προωθήσουμε πριν ε, προωθήσουμε ε, τους γεωπολιτικούς μας στόχους. Μόνο εάν επιτύχουμε τους στόχους μας, τους γεωπολιτικούς, μόνο τότε είναι δυνατόν να έχουμε αρκετή ισχύ, ειδικό βάρος, τέλος πάντων, τόσο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τις αρχές μας. Και βάζω τελεία λέγοντας ότι ίσως ο κύριο Μπέλντερ θα μπορούσε να δει τι άλλες ε, σημαντικέ τροπολογίε μπορεί να κλείσει, γιατί όντω υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίε, ε, έχω και εγώ κάποιε διατάξει να προτείνω, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε και σε και τώρα. Κύριε Μπέλτερ, για να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και την καλή συνεργασία τον κύριο Κασουλίδη, τον κύριο Coffer και τους υπόλοιπους, τον κύριο Τάνοκ, τους υπόλοιπους συναδέλφους. Συνοψίζοντας, αντιλαμβάνομαι πως η συμβαστική τροπολογία 10 ε, η αρχική διατύπωση εκεί πέρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα υπόλοιπα, εντάξει, ε, προφανώς ε, αναφέρει την αποδοχή από την κοινωνία κτλ. Και τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν την θέση της Ταϊβάν. Είμαι περίεργος για το πώς θα κυλήσουν οι διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των ομάδων και τις επόμενες ημέρες ε, θα αναλογιστώ το ζήτημα, όπως είπα, της συμβαστικής τροπολογίας 10 ε, ε, και της Ταϊβάν, όπως είπε και η κυρία Κοπάιν, μια εξόχως περίπλοκη έκθεση. Αλλά βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια πράγματα όπως είπε και ο πρόεδρος τα οποία βρίσκονται εκτός ε, του πεδίου της ε, έκθεσης η πνευματική ιδιοκτησία και τα λοιπά δεν είναι το αντικείμενο της έκθεσης αυτής. Τέλος, κύριε Σεβερίν, είδα τις τροπολογίες σας, αλλά Ε, οπότε φαίνεται θέλουν να ανοίξουν μια μεγάλη πολιτική συζήτηση και δεν λαμβάνουν μια συγκεκριμένη πολιτική θέση και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα μου εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, να σκεφτούμε, αλλά δεν μπορούν να μπουν αυτά τα πράγματα εντός της έκθεσης. Ε, οπότε για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στην έκθεση αυτή δεν βλέπω ακριβώς την χρησιμότητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους ε, τώρα όσον αφορά τις συζητήσεις για την Ταϊβάν και το Κομμουνιστικό Κόμμα όπως σας είπα θα τα ξαναδούμε τα ζητήματα οπωσδήποτε πριν ε, πάμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλντερ για την δουλειά σας. Ε, τελειώνουμε με αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξης και πάμε κατευθείαν στο επόμενο, το οποίο είναι εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ. Ξεκινάμε με τον ε, εισηγητή, τον κύριο Μαύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να θυμίσω ότι το ψήφισμα συνοδεύει το κείμενο του PCI. Και νομίζω πως από αυτή την οπτική θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τις ε, τροπολογίες. Η δική μου αξιολόγηση του PCI είναι θετική. Πιστεύω δηλαδή πως αυτό το μέσο είναι κατάλληλο για να ευνοηθεί η πορεία προς τον εκδημοκρατισμό της ζωής και της κοινωνίας του Ιράκ, συμβάλλοντας αντικειμενικά στην υπέρβαση των πολιτικών εμποδίων που ακόμα καλανίζουν τη ζωή αυτών των χωρών και έπειτα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα χρήσιμο μέσο για να βοηθηθεί το Ιράκ. Από αυτήν την άποψη αξιολόγηση που κάνω για τις 132 τροπολογίες που υποβλήθηκαν ε, αυτή την οπτική ακολουθούν. Δηλαδή να μην ε, να κάνουμε κριτικές για το Ιράκ, να πούμε για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση, αν σέβονται τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτική κρίση, αν μπορούν να μπορέσει τελικά το Ιράκ να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία διανύει, αλλά όλα αυτά σχετίζονται με το PCI και άρα δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε μια θετική κατέθεση σε σχέση με τις αξίες αυτού του κειμένου. Και γι' αυτό το λόγο στη συνεδρίαση που θα γίνει σήμερα με τους σκιώδεις εισηγητές στις 2 με 3 και που γίνεται έτσι σύντομα γιατί μετά εγώ πρέπει να ακολουθήσω την αντιπροσωπεία της Ένωσης με τις ε, ΙΠΑ σε μια αποστολή που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Ουάσιγκτον. Θα μπορέσουμε λοιπόν έτσι να αντιμετωπίσουμε τις ε, αντιφάσεις μέσω των συμβιβαστικών τροπολογιών. Θα μπορέσουμε δηλαδή εύκολα να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να μειώσουμε τον αριθμό των ε, τροπολογιών. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες ε, ε, λάβαμε πολλά στοιχεία από την κοινωνία των πολιτών του Ιράκ, από πολλούς φορείς ε, που θέλησαν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι όλο το κείμενο του ψηφίσματος ε, έχει συνταχθεί με συμμετοχή πολλών συναδέλφων που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να εκφραστεί η γνώμη του Κοινοβουλίου στα, για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράκ. Εγώ είμαι πεπισμένος για την ποιότητα πολλών από τις τροπολογίες που μου υποβλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάουρο και τώρα ξεκινάμε με τους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Καταρχήν η κυρία Κοπά. στην πρώτη συζήτηση που κάναμε φάνηκε ότι υπάρχει κοινό τόπος ε, με τον συνάδελφο Μάουρο σχετικά με την έκθεσή του και πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητη η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ. Αρχικά γιατί είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε ουσιαστικά τη χώρα αυτή στο μακρύ δρόμο προς την ομαλότητα και τη σταθεροποίηση αλλά και δεύτερο γιατί η βία και η τρομοκρατία που ταλαιπωρούν τη χώρα μπορούν να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά μόνο μέσα από την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας. Μέσα από τη Συμφωνία είμαστε σε θέση να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών και θεωρώ πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο ότι η Συμφωνία περιλαμβάνει δική ρήτρα για την προσχώρηση του Ιράκ στο ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι επίση σαφέ ότι αν το Ιράκ δεν κατορθώσει να κάνει πρόοδο στον πολύ ευαίσθητο αυτό τομέα, τότε τα προγράμματα συνεργασίας και ανάπτυξης θα επηρεαστούν ουσιαστικά. Ε, στην έκθεση του συναδέλφου Μάουρο έχουν κατατεθεί 132 τροπολογίες. Ε, μερικές από αυτές αναφέρονται στην περίοδο του πολέμου ε, πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση που αν θέλουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε το Ιράκ πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και όχι πίσω. Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος κατέστρεψε αυτή τη χώρα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να συνεχιστεί πολιτική διαδικασία και να γίνουν εκείνες οι ενέργειες ώστε να παγιωθεί η δημοκρατία και να σταθεροποιηθεί το καθεστώς. Πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε όλες τις τροπολογίες που τονίζουν την εθνική συμφιλίωση, την εθνική συνοχή, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, που καταδικάζουν τη θρησκευτική βία προς όλες τις κοινότητες, τις τροπολογίες που αναφέρονται στις γενικευμένες παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κατάργηση της θανατικής ποινής και φυσικά στην ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας. Το Ιράκ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια χώρα που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο της ασφάλειας, της ενέργειας, της οικονομίας. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον μας να καταστεί το γρηγορότερο δυνατό περιφερειακός παίκτη και ένας αξιόπιστος διεθνής εταίρος. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάθε λόγο να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ε, δεν είχα την ευκαιρία να συμβουλευτώ τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν προταθεί. Έχουμε τη συνάντηση σήμερα, οπότε επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ την επόμενη, στην επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, e Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοπά. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τάνοκ για την ECR. Δεν ζήτησα το λόγο ναι, εμένα, αλλά ευχαρίστως να πω δύο λόγια. Καταρχήν να συγχαρώ τον Μάριο Μάουρο για την έκθεσή του. Προφανώς το Ιράκ ε, αποτελεί ακόμα μια πρόκληση και ε, καλωσορίζω τον ορισμό της, του επικεφαλής ε, Γιάννη Μπάσκοβα της αντιπροσωπείας της Ένωσης που παρετήθη, συγγνώμη, που μένει στην Βρετανική Πρεσβεία. Εγώ από παλιά που υποστήριζα τους χριστιανούς του Ιράκ και της Συρίας πιστεύω πως δεν γίνονται αρκετά πράγματα ε, για να προστατευθούν. Πολλοί από αυτούς έχουν ε, προσφύγει στη Συρία, έχουν καταφύγει στη Συρία που πάλι θα πρέπει να φύγουν γιατί είναι μια μειονότητα η οποία διώκεται πολύ έντονα Ανησυχώ ιδιαίτερα επίσης για τη στήριξη που δείχνει ο Αλμαλίκη σε ένα είδος ε, εκπροσώπησης του Ιράν στον Αραβικό Σύνδεσμο και φαίνεται να στηρίζει τα όσα συμβαίνουν στη Δαμασκό και επιτρέπει την υπέρπτυση των Ιρανικών ε, φορτίων όπλων. Ε, αυτά δεν αναφέρονται όμως στην έκθεση, παρότι την έψαξα. Τι αναφέρεται, δεν το είδα, δεν το είδα. Μόλις την είδα και την ε, είδα έτσι στα πεταχτά. Αλλά όπως σας είπα, ούτως ή άλλως είναι πρόκληση το Ιράκ. Πρέπει να στηρίξουμε την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη, την περαιτέρω οικοδόμηση και να, συγχαρούμε, και να συγχαρούμε για την ειρήνη και τη σταθερότητα της οποίας χαίρει η κουρδική αυτόνομη δημοκρατία στο βόρειο Ιράκ. Είχα επαφές με τους εκπροσώπους τους στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο. Κατά τα άλλα, να πω και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Μάουρο και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Ιράκ με μένα ενδιαφέρον, γιατί πολλή δουλειά ακόμα πρέπει να γίνει, <laughs> ώστε να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη δημοκρατία και την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. One minute, please. Κύριε Γκόμες, για ένα λεπτό. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάουρο ε, πολύ σημαντικό το κείμενο. Και η συμφωνία μπορεί όντω να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πράγματα, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα έχει τα μέσα επιτόπου και την αυτονομία από να μπορεί να κινηθεί και να δουλέψει. Προσπάθησα εδώ να τοποθετήσω μια προοπτική που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει λάθος αντιληπτή στο Ιράκ, ότι δηλαδή θέλουμε να μεριμνήσουμε για τις χριστιανικές κοινότητες. Έχουν αποτελέσει στόχο και θα ήταν μεγάλη απώλεια για το Ιράκ να χάσει αυτή την πολυμορφία που δίνει η χριστιανική κοινότητα και άλλες κοινότητες στη χώρα κατά τη διάρκεια των αιώνων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας απασχολεί μόνο το θέμα των χριστιανών, εφόσον και άλλες, πλειοψηφ... και άλλες κοινότητες όπως οι Σιήτες και οι Σουνίτες έχουν υποφέρει τόσο πολύ και εξακολουθούν να υποφέρουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τρομοκρατικές επιθέσεις. Οποιοδήποτε άνθρωπο είτε είναι χριστιανό είτε είναι μουσουλμάνος, συμπάσχει. Νομίζω Το θέμα του ΜΚΟ θα πρέπει να παραμείνει στο Ιράν και όχι στο Ιράκ. Θα πρέπει να αφήσουμε τη συνεργασία μας με το Ιράκ να ε, πνιγεί από, τη συνεργασία, από το, την ατζέντα του ΜΚΟ και δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ε, αφήνουν να συμβεί αυτό. Συμφωνώ με την ε, κυρία Κοπά ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε υψηλές προδιαγραφές από το Ιράκ όσον αφορά τους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε ακόμα δύο-τρεις παρεμβάσεις και ο Αμερικανός πρέσβης περιμένει ήδη. Γι' αυτό δίνω ένα λεπτό στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχα την ευκαιρία να σας εξηγήσω τι πρεσβεύει η πολιτική μας ομάδα. Θεωρώ ότι κάποια κράτη-μέλη ξεκίνησαν πόλεμο, πόλεμο παράνομο, προληπτικό, βασισμένο σε ψέματα. Και το μόνο το οποίο ήταν σίγουρο είναι ότι ωφέλησαν το, τον υπουργό τους που ασχολείται με. Ή τόσο βοήθησαν την, την, την προμήθεια σε πετρέλαιο. Οπότε ε, είπαμε την ανάμεξη του ΟΗΕ, αλλά είχαμε τόσες, τόσες δεκάδες χιλιάδων να, να σκοτώνονται και 70.000 επίσης Αμερικανοί ε, ε, σκοτώθηκαν σε αυτήν την παρανομή εισβολή, απερίμωση, οι άλλες όπως είπε η κυρία Ιβάσκοβα στην τελευταία έκθεση όσον αφορά το Ιράκ και εκεί πέρα μας έχει περιγράψει μια πραγματικότητα 99% του, του Ιράκ μαστίζεται από φτώχεια, δεν έχει δικαιοσύνη, δεν έχει ασφάλεια. Εκατοντάδε χιλιάδε είναι, είναι οι πρόσφυγε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαόρο για την έκθεσή του. Νομίζω ότι έχει καλύψει και μια δικιά μα τροπολογία. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό, γιατί αν πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία σύνθεσης είναι για να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγγνώμη για, για αυτή την, την διάλυση, την ερήμωση που ποτέ δεν έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάγερ. Κύριο Λαντσμπέργκης τώρα για ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ασχοληθώ μόνο με τον παράγραφο 9. Προτείνουμε εδώ πέρα στήριξη από τον κύριο Στίβενσον, αλλά αν δεν περάσει υπάρχει δική μου η διόρθωση στο κείμενο. Η νέα διατύπωση λοιπόν της παραγράφου 9 θα έχει ως εξής. Το Κοινοβούλιο επικροτεί την δέσμευση των Ιρακινών αρχών να εξασφαλίσουν τις ε, επαρκείς συνθήκες διαβίωσης ε, και θανάτου για τους 50 κρατούμενους στο στρατόπεδο Άστραφ. Ζητάει από τις ΗΠΑ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επανεγκατάσταση ή επαναπατρισμό σε ένα δημοκρατικό Ιράν. Χρειάζεται αυτό. Των κατοίκων του στρατοπέδου ε, αυτού έτσι ώστε να βρεθεί μια οριστική λύση για τους κρατούμενους αυτούς στην Ιρακινή επικράτεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαντσμπέργκης, ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ τη δουλειά του κύριου Μάουρο. Εγώ στήριξα πολλές ε, τροπολογίες που αναφέρουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτιμώ πως κάποια ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν συμπεριληφθεί και θα ήθελα να τονίσω πως υπάρχουν πολύ περισσότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, έχω σοβαρές ανησυχίες για το πρόβλημα των Ιρανών προσφύγων που πήγαν από το στρατόπεδο Άστραφ στο στρατόπεδο Λίμπερτι. Παρακολουθώ το ζήτημα εδώ και λίγο καιρό και δεν ε, συμφωνώ με τον θετικό τόνο της αρχικής παραγράφου 9. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες η κατάσταση εκεί είναι πολύ πιο δραματική και χρειάζεται την άμεση προσοχή μας και συνεισφορά μας στην λύση με τρόπο γρήγορο, σεβόμενοι πλήρως τα βασικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κούπαν. Για να συνοψίσει ο κύριος Μάριο Μαουρό. Μάλιστα, Πρόεδρε, σε μερικά δευτερόλεπτα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και για τα καλά τους λόγια. δεν υπάρχει καμιά κανένα πρόβλημα να αναφέρουμε και να καταγγείλουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορούμε όλα αυτά να τα τοποθετήσουμε σε μια θετική οπτική που σχετίζεται με την φύση του PCI, μια συμφωνία δηλαδή που θα επιτρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα στο Ιράκ να φύγει, να βγει από την κρίση του που αντιμετωπίζει ως κράτος και ως έθνος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάουρο. Μπορούμε να κλείσουμε. να καλωσορίσουμε τον Αμερικανό πρέσβη. Έχω τώρα λοιπόν την τιμή να καλωσορίσω τον πρέσβη Κέναρτ ε, στην Επιτροπή μας. Ειδικά τώρα μετά τις ε, Αμερικανικές εκλογές. Και την εκλογή, επανεκλογή του Πρόεδρου. Και στη θέση λοιπόν του Πρόεδρου του παραδοσιακού μας εταίρου, τον είπα. Δίνω τον λόγο λοιπόν στον ε, κύριο Πρέσβη, τον κύριο Κένερτ να ξεκινήσουμε λοιπόν με την δική σας εισαγωγή και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια των βουλευτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι νομίζω μια πολύ καλή εποχή για να συναντηθούμε καθώς ε, όπως πολύ καλά ξέρετε είχαμε την επανεκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα αλλά είναι και σημαντική εβδομάδα στην ε, Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Σούλτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει συναντήσει στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο Μπάιντεν και άλλα στελέχη της κυβέρνησής μας και αναμένουμε τον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο που θα ξεκινήσει την Ουάσιγκτον την ε, Παρασκευή. Είναι λοιπόν σημαντική η εβδομάδα. Δεδομένης επανεκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα είναι μια σημαντική στιγμή για εμάς για να συναντηθούμε, να δούμε τα της σχέσεώς μας και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασχολήθηκαν με τις εκλογές μας. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που είδα προεδρικές εκλογές εκτός των ΗΠΑ. Και ήταν φοβερό το πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος για την πολιτική της χώρας μας. Και τώρα ο κόσμος αναρωτιέται το τι σημαίνει αυτό, πώς θα είναι η δεύτερη θητεία του Προέδρου για τη ΣΥΠΑ και για τον κόσμο. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανέλαβε την εξουσία αποδεχόμενος βεβαίως ε, και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ενός πολύ πιο διασυνδεδεμένου κόσμου στον 21ο αιώνα και είπε πως η συνεργασία μεταξύ των ε, χωρών δεν είναι ε, επιλογή είναι ο μόνος τρόπος για να προωθήσουμε αυτά τα οποία μας απασχολούν ως ανθρωπότητα και είναι νομίζω σαφές τώρα πως στην πρώτη του θητεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια τήρησε την δέσμευσή του για να έχουμε ξανά σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, με πολυμερείς οργανισμούς και ειδικά τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να αναγνωρίζετε πως έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν για να έχουμε βαθύτερες επαφές με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα από την πολύ παραγωγική σχέση εργασίας που έχουμε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Βεβαίω, όπως πάντα, υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, αλλά καθώς κάνουμε έναν απολογισμό της πρώτης θητείας του Προέδρου, πρέπει να σας πω πως η κυβέρνησή μου έχει ωφεληθεί πάρα πολύ από την ε, αυξημένη επαφή που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαμε, αυτό αποτελεί θεμελιολήθεια της πολιτικής μας και σε όλα τα επίπεδα ερχόμαστε σε επαφή με τους ομολόγου μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επενδύσουμε σε μια ουσιαστική για εμά σχέση. Είχαμε λοιπόν μια ξεκάθαρη επιλογή ως Αμερικανικός λαός και ο Αμερικανικός λαός επέλεξε με τρόπο φασιστικό να διατηρήσει τον πρόεδρο Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, το όραμα του πρόεδρου συμπεριλαμβάνει τη δουλειά που είναι η συνεργασία μαζί σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για εμάς εκπληκτικό το ότι στην πρώτη θητεία του Προέδρου Ομπάμα είχαμε κοινέ προτεραιότητες στην εξωτερική πολιτική και αναμένουμε αυτό να συνεχίσει και στη δεύτερη θητεία. Βεβαίω, η συνεργασία μας είναι ευρύτατη και βαθύτατη. Εγώ βρισκόμαι στο κέντρο αυτής της σχέσης μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε μέρα που περνάει Εκατοντάδε ζητήματα αποτελούν αντικείμενο εργασία σε όλα τα επίπεδα τη κυβέρνησή μα και για να τα συνοψίσω εντάσσονται σε τέσσερι κύριε κατηγορίε. Πρώτον, προσπαθούμε να στηρίξουμε τι φιλοδοξίε των ανθρώπων σε νέε δημοκρατίε. Δεύτερον, η δουλειά που κάνουμε για τι παγκόσμιε απειλέ ιδιαίτερα την τρομοκρατία. Τρίτον, συντονισμός ε, της βοήθειάς μας στους πιο ευάλωτους του κόσμου και τέταρτον με τρόπους για να αυξήσουμε την οικονομική και αριθμιστική συνεργασία μας. Θα μιλήσω τώρα σύντομα για αυτά τα οποία κάνουμε σε κάθε ένα από αυτούς τους τέσσερις τομείς. Θεωρούμε πως η στήριξη των φιλοδοξιών των ανθρώπων στις νέες δημοκρατίες ε, είναι η σημαντικότερη δουλειά που κάνουμε από κοινού. Έχουμε ήδη ε, ένα δημοκρατικό μέλλον που διαφαίνεται στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην περιοχή αυτή, στη Λιβύη, τη Συρία, Αίγυπτο, την Ισία κτλ. Και αυτό θα συνεχιστεί. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΙΠΑ καλώς όρισαν ε, την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολούθησε με μεγάλη ανησυχία, αλλά αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε μία περίοδο σχετικής ηρεμίας και βεβαίως καταλήξαμε σε αυτή την συνεννόηση μετά από διπλωματικές προσπάθειες Αιγύπτου, Ισραήλ, των Παλαιστινιακών Αρχών, των λοιπόν στην περιοχή, του ΟΗΕ, βεβαίως των Ευρωπαίων Συμμάχων μας. Όπως είπε η υπουργό η κυρία Κλίντον την προηγούμενη εβδομάδα, είναι κρίσιμη η στιγμή αυτή για την περιοχή και βέβαιως ο κόσμος αξίζει να ζει χωρίς ε, φόβο βίας. Τώρα θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα διαρκές αποτέλεσμα το οποίο θα προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα και την αξιοπρέπεια και τις φιλοδοξίες Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με του εταίρου μα στην περιοχή για να βελτιωθούν οι συνθήκε για του ανθρώπου στην Γάζα και για να υπάρχει ασφάλεια για το λαό του Ισραήλ. Τέλο, κάθε βήμα πρέπει να μα πηγαίνει πιο κοντά σε μια συνολική ειρήνη για όλου του ανθρώπου τη περιοχή. Στηρίζουμε τη δημιουργία ενό Παλαιστινιακού κράτου στο πλαίσιο μια λύση δύο κρατών ω αποτέλεσμα άμεσων συνομιλιών χωρί ε, προαπαιτούμενα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ξεκολουθούμε να είμαστε κατά των Παλαιστινιακών προσπαθειών για αναβάθμιση του καθεστώτος του στον ΟΗΕ εκτός του πλαισίου μια συμφωνημένη λύση. Για να στραφώ σε άλλου τομεί το Ιράν Χαρήκαμε για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένει με το βραβείο Ζαχάροφ σε δύο θαραλέους αντιφρονούντες και συγχαίρουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο Αφγανιστάν. Εμεί και οι διεθνεί μα εταίροι προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την πολιτική και την οικονομική μετάβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε μια μετάβαση στο τέλο του 2014 και θα έχει κρίσιμη σημασία για τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του εταίρου μα να στηρίξουν τι αφγανικέ δυνάμει ασφαλεία για να ε, παρέχουν ασφάλεια και να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Καλωσορίζουμε επίσης ε, την ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση και την ένταξη του Αφγανιστάν στα περιφερειακά όργανα της Κεντρικής Ασίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά για τα ζητήματα Βαλκανίων. Η Υπουργό, η κυρία Κλίντον και η Πατικπρόσωπος, η ε, κυρία Άστον, συνεργάστηκαν σχεδόν τέλεια σε Βοσνία, Σερβία, Κοσφοπέδια για να ενθαρρύνουν τους ηγέτες να ξεπεράσουν ε, τις εθνοτικές διαφορές και να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις που ζητάνε οι πολίτες τους. Επίσης συνεργαστήκαμε στην Ουκρανία, θα είδατε πρόσφατα, πως η Κάθη και η Χίλαρη Κλίντον ε, συνέταξαν από κοινού ένα άρθρο στις εφημερίδες ε, και ζητούν από τις Ουκρανικές αρχές να γίνουν οι εκλογέ με τρόπο ελεύθερο και δίκαιο. Επίση, συνεργαζόμαστε στενά στη Λευκορωσία. Υπάρχει δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Στην Ασία. Βλέπουμε ιστορικές ανακατατάξεις στη Γερμανία. Έχουμε συνεργαστεί και πάλι στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε επισκέψεις πολύ υψηλού επίπεδου από την κάθε άστον τη Χίλαρη Κλίντον και προσφάτως ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε την πρώτη του επίσκεψη στη Βυρμανία όπως έκανε και ο πρόεδρος Μπαρόζο. Άλλωστε όλες αυτές οι επισκέψεις τονίζουν τις κοινές μας προσπάθειες για να στηρίξουμε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη χώρα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πάρα πολύ βασικό το ότι τώρα ο Σταύρο Τζαμπενίδη, ο πρώην ε, Ευρωβουλευτή, έχει γίνει τώρα ειδικό απεσταλμένο για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και πολλοί από εμά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ε, στένα με τον Σταύρο και ξέρω ότι πρόκειται την την, την, την ευφυΐα του, την εμπειρία του, όλα αυτά να τα μεταλαμβαδεύσει να τα χρησιμοποιήσει στη, στη θέση και επίσης έχουν γίνει συναντήσεις με επίσημες πηγέ στη, στην Ουάσιγκτον και οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα θα αποτεθούν καλύτερα παντού στον κόσμο και θα προηθούν τα δικαιώματα των γυναικών αλλά των ε, ομοφυλοφίλων λεσβιών κλπ. Σε, σε όλο τον κόσμο και τώρα να δούμε τι θα γίνει με τι παγκόσμιε απειλέ και την τρομοκρατία όπως όλοι γνωρίζετε, ότι ε, αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα για μας. Και συνεχίζουμε το να συνεργαζόμεθα όσον αφορά την, την, την τρομοκρατία, την μη διάδοση των πυρηνικών, την αστάθεια που βοηθά ε, την τρομοκρατία. Τα τελευταία χρόνια επίσης πάρα πολύ στενά δουλέψαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα εκείνα. Και επίσης ε, θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μας για το PNR αλλά και για την αναζήτηση των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για όσα κάναμε σε σχέση με, την, με τη φόρτωση των αεροπλάνων, με την ασφάλεια στα αεροδρόμια, για το, το PNR, για το TFTP, για το SWIFT. Όλα αυτά ξέρουμε πόσο σας εδίχασαν εδώ, πόσο ήταν αμφιλεγόμενα και πάντως δεν μπορούμε παρά να σας συγχαρούμε για το έργο το οποίο επιτελέσατε και είμαστε ευγνώμονες ε, για την υποστήριξή σας. Και πέρσι επίσης είχαμε το φόρουμ κατά της τρομοκρατίας και ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργαστήκαμε ε, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, απειλές προς και εμάς και προς άλλες χώρες. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο τώρα είπαμε ότι έχουμε στην Τινησία ε, <clears throat> το κέντρο κατάρτισης για το διεθνές δίκαιο και επίσης αυτό πρόκειται να εκπαιδεύσει κόσμο από την Ισία και Μέση Ανατολή. Η Λιβύη βέβαια τα τελευταία χρόνια απασχόλησε τα πρώτα σέλιδα και συνεργαστήκαμε και σε αυτό μέσα όσον αφορά τις κυρώσεις τόσο ώστε τελικά να γονατίσουμε το καθεστώς Καντάφη ε, το προσεκά του στοιχεία, τις εξαγωγές του πετρελίου, τα, τα παγώσαμε και όσον αφορά τις κυρώσεις ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί εκτός από τη Λιβύη και εις βάρος του Ιράν. Ε, συντονιστήκαμε πάρα πολύ συχνά, στενά με, την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω είναι σαφές ότι οι κυρώσεις εκείνες ε, τις οποίες ε, επιβάλαμε από κοινού βοήθησαν το να ξανακαθίσει το τραπέζι των το Ιράν και να συνομιλήσει με την κοινότητα. Με την καθιάστα να συνεργαζόμαστε με το επιτελείο της για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, βοηθούν στην μη διάδοση των οικονομικών της καταστροφής για την ε, Βόρεια Κορέα και καλούμε ε, την χώρα αυτή να κάνει το καθήκον της όσον αφορά τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Στο Σαχάλ, επίσης, στο Σαχέλ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις τρομοκρατικές απειλές και επίσης έχουμε κάποιες σχετικές εξελίξεις στο βόρειο τμήμα του Μαλή. Και επίσης είναι αλήθεια ότι εκεί η κατάσταση ε, επιβάλλεται να έχει μια περιφερειακή λύση. Έχουμε εκεί πέρα ε, την πολυεθνική δύναμη με ηγεσία αφρικανική και έτσι βοηθούμε την κυβέρνηση ε, του Μάλι να αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες. Τώρα όσον αφορά την ανάπτυξη. Ε, ενδιαφέρον στοιχείο της εταιρικής μας σχέσης είναι ότι όλα όσα γίνονται είτε είναι ανθρωπιστική κρίση, είτε είναι οποιαδήποτε κρίση, ε, συνεργαζόμαστε. Τον Απρίλιο οργανώσαμε αυτή την διάσκεψη των δωρητών στο Ναϊρόμπι. 1,2 δισεκατομμύρια ε, ελκύσαμε ως ενίσχυση ε, των Αφρικανών στο κέρας Αφρικής και στο Σαχέλ. Στον Ναϊρόμπι επίσης ε, συνεχίστηκε η συνάντηση για να δούμε πώς ήταν πιο αποτελεσματικά τα προγράμματά μας. Επίσης κάνουμε ό,τι πρέπει να το χέρι μας τόσο ώστε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια προς την ε, Συρία για την εκεί κρίση. 65.000 ε, δολάρια διαθέσαμε για την Συρία, δηλαδή 75% του συνόλου των όσων έδωσαν ε, όλοι οι δωρητές για την κρίση στη Συρία. Εσείς και εμείς τα δώσαμε αυτά. Τώρα, θέλω να ολοκληρώσω για κάτι το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με την ε, εξωτερική πολιτική, αλλά αφορά την συνεργασία μας όσον αφορά τα οικονομικά και όσον αφορά την νομοθετική πολιτική, ότι, ότι χρειάζεται να έχουμε αποτελεσματική, οποιαδήποτε χώρα χρειάζεται αποτελεσματική εξωτερική πολιτική όσον αφορά την ενίσχυση έτσι της οικονομίας, γιατί ε, ε, είχε χτυπηθεί και η δική σας και η δική μας οικονομία από αυτή την ε, πιο σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση, τη μεγαλύτερη από την, εποχή του κράχ, οπότε θα πρέπει και εδώ να δούμε πώς μέσω της συνεργασίας μας θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη η οικονομική εταιρική μας σχέση είναι πιο σημαντική παγκοσμίω. Και εκπροσωπεί ένα τρεις δολάρια εμπορίου. Αλλά αν συνδυάσετε και τις ε, επενδύσεις ε, εξωτερικές θα πάμε για τεσσερα 3 Οπότε δεν μπορεί κανείς παρά να δεχθεί ότι παρά όμως τη μεγάλη μας αυτή επιτυχία έχουμε ακόμα πολύ έδαφο για βελτίωση των επιδόσεων. Οπότε να δούμε πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε, πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή μας την συνεργασία. Και τρία χρόνια που έχω αυτή τη θέση δεν έχω δει πιο, πιο, πιο καλό κλίμα ε, για να πάνε τα πράγματα καλύτερα και αυτό οφείλεται σε εσά εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε και τώρα έχουμε σημαντικές επαφές σε αυτό που ονομάζουμε ομάδα υψηλού επίπεδου για ανάπτυξη και θέση εργασίας. Θα γίνουν επίσης σημαντικές επαφές και στην Ουάσιγκτον για το ίδιο θέμα και επίσης θα γίνει αυτό όσον αφορά την, τον διάλογο τον ε, ε, διατλαντικό που αφορά τους συνομοθέτες και έτσι θα δούμε πώ θα ξενεθούν και άλλε ευκαιρίε στους επόμενου μήνε. Τώρα όσον αφορά την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Αυτό έχει σχέση με το PNR, το TFTP και την εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων εδώ. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε και θα πρέπει να ε, επικαιροποιήσουμε ε, και να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας. Και εσείς εδώ, όσον αφορά τα εμπορικά δεδομένα, ε, ε, δουλεύετε και άρα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε κάποια συστήματα που εντάξει, να μην είναι ε, ταυτόσιμα, να μην είναι τέλεια, αλλά τέλο πάντων είναι συμβατά. Οπότε, όσον αφορά τη δεύτερη θητεία Ομπάμα, είναι σημαντικό το έργο το οποίο αρχίσαμε κατά την πρώτη θητεία Ομπάμα πρέπει και να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί όπως ε, μας έδειξαν τα εντυπωσιακά δραματικά παγκόσμια γεγονότα, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις και που είναι πιεστικές και όπως είπε και ο πρόεδρος των πριν από μερικές εβδομάδες, είπε ότι αρχίζει πιο αποφασιστικά τη δεύτερη θητεία. Μεγαλύτερη έμπνευση, μεγαλύτερη όρεξη για το έργο που έχει επιτελέσει, οπότε και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, όπως έγινε ακριβώς και στην πρώτη θητεία. Στενή συνεργασία θα γίνει πάλι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευράς ε, της διοίκησής μας, κυβέρνησής μας, του Υπουργείου μας, ξέρουμε ότι ο πιο καλός μας εταίρος για αυτές τις προκλήσεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδείχθηκε στο παρελθόν. Σας συγχαίρομαι για το βραβείο Νόμπελ και γνωρίζουμε ότι αυτό συμβολίζει όχι μόνο το έργο το έργο σας του παρελθόντος, αλλά και το τι θα κάνετε. Ελπίζουμε σε συνεργασία μαζί μας, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είσαστε ο πιο σημαντικός μας σύμμαχος όσον αφορά την ευημερία και την ειρήνη που θέλουμε να προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο. Thank you very much, Ambassador Kenneth. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παζευτά. Όντω είναι μακρύ ο κατάλογο των θεμάτων συνεργασία μεταξύ ημών και ημών και θεωρούμε και εμείς ότι εσείς είστε ο πιο σημαντικός στρατηγικός μας εταίρος, τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και επίσης τα διμερή ζητήματα. Τώρα, να κάνουμε δύο γύρους παρεμβάσεων των συνάδελφων εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ξεκινούμε με δίλεπτες ε, παρεμβάσεις από τους συντονιστές. Πρώτα-πρώτα για το ΕΛΚ, ο κύριος Σαλαφράγκα. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά, κύριε Κέναρντ για την συνεργασία σας, για την ε, συνεχή σας παρουσία σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου μας. Νομίζω ότι πάρα πολύ καλά τα είπατε όσον αφορά το, το, πόσο είναι συντονισμένη στην εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η ΕΠΑ. Και εσείς από τις θέσεις σας νομίζω μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και ε, είπαμε ότι ε, πρέπει να αντιμετωπίσετε με Μέση Ανατολή, Αίγυπτο, ε, Αραβική Άνοιξη. Ε, όλα αυτά αξίζουν την προσοχή σας, οπότε παρακαλώ πέστε μας κύριε Πρέσβη. Το Κοινοβούλιο, ξέρετε, την περσμένη εβδομάδα έγινε ένα ψήφισμα όσον αφορά τη σύγκρουση στην Γάζα και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ θετική η παρουσία της, ε, τον είπα, στην ε, περιοχή και ήταν σημαντική συμβολή όσον αφορά την ε, κατάβευση του πυρός και οπότε θα δούμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με την Παλαιστίνη και τον ΟΗΕ το καθεστώς δηλαδή που θα, έχει η Παλαιστίνη τελικά τα πράγματα είναι αβέβαια ο Ιησούς αποσυρθεί από, από τη θέση ε, από το να βοηθά, τέλος πάντων αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τη Παλαιστινική αρχή Τι λέτε εσεί. Τι λέτε ότι μπορεί να γίνει ε, όσον αφορά την Παλαιστίνη και τον ΟΗΕ. Τώρα κάτι άλλο για την Κίνα και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κλιμάκωση, την αποκλιμάκωση μάλλον της έντασης στη θάλασσα της Κίνας. Το Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, ξανακάθισε τον Τραπεζικό Παντέσιο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνεχίζεται ο διάλογος που Κούβα. Ε, και εσείς και εμεί θέλουμε εκεί πέρα να δούμε πώ θα γίνει δημοκρατικός μετασχηματισμό και γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο της Ένωσης ε, παγίω ζήτησε ε, από ε, την εξωτερική υπηρεσία της Ένωσης να προχωρήσει στο να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία και Είπαμε ότι τώρα, τώρα που τέλο πάντων ξεμπέρδεψε με τα ο, ο πρόεδρος Ομπάμα, τώρα μπορεί να είναι πιο ευέλικτο όσον αφορά την ε, Κούβα. Ευχαριστούμε κύριε ε, Σαραφράγκα και τώρα για του Σοσιαλιστέ Δύο λεπτά η κυρία Γκόμες. Ε, ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε Πρέζη. Χάρηκα και ανακουφίστηκα που επανεξελέγει ο πρόεδρος Ομπάμα, ειδικά όσον αφορά την προοδευτική αφήγηση για την οικονομική κρίση, αντίθεση, σε αντίθεση με όσο συμβαίνουν στην Ευρώπη, με την ε, προσέγγιση της λιτότητας η οποία χειροτερεύει τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα σχόλια του συναδελφού σας Φράγκα για την ε, κατάβαση του πυρός στη Γάζα. Το εάν θα στηρίζεται μια αποπερινικοποιημένη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπιστούν οι φοβερέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, δηλαδή ο εξοπλιστικός ε, αγώνας που έχει ξεκινήσει με αφορμή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για τις παγκόσμιες ε, απειλές. Πώς βλέπετε την αύξηση της στρατιωτικής ισχύως της ε, Κίνας με τρόπο αδιαφανή. Και μιλήσατε για παγκόσμιες απειλές και συγκεκριμένα το Σαχέλ και ειδικά το Μαλί. Αλλά η ΕΠΑ ΕΕ ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την ε, βάση του Λάζες ε, στο μέσον του Ατλαντικού και μάλλον λόγω λιτότητας οι Κινέζοι λένε πως θέλουν αυτοί τώρα να πάρουν την θέση των ΙΠΑ στη βάση αυτή. Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν αυτές τις στρατηγικές προκλήσεις η ε, χώρα σας. Τέλος, να σου ρωτήσω το εξής. Δεν δέχομαι ε, τα περί εξαιρετικής θέσης των ΙΠΑ για την δικαιολόγηση των εκτελέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πότε θα συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση Ομπάμα πως ε, κάτι τέτοιο θα πλήξει τη ΣΥΠΑ εάν συνεχιστεί, ε, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε, κύριε Κυρία Νέιτς για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη. Καλώς ήρθατε. Και θα ήθελα και εγώ να πω πως είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όταν μάθαμε πως ο Αμερικανικός λαός αποφάσισε να επανεξελέξει τον Ομπάμα. Μια σωστή απόφαση εκατομμυρίων Αμερικανών. Σαν όπως και άλλοι συνάδελφοι, εγώ ήμουν στην Σαρλότ, στο συνέδριο των Δημοκρατικών και αρνητικές, ε, μια αρνητική εμπειρία που είχα ήταν το ότι συνειδητοποίησα το πόσο λίγο ανέφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση. European States. Ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβάνομαι πως το συνέδριο είναι εσωτερική υπόθεση. Και βεβαίως ε, απευθύνεται στον Αμερικανικό λαό τους ε, ψηφοφόρους των δημοκρατικών ε, πρώτα απ' όλα και μετά το κοινό, το ευρύτερο. Αλλά οπωσδήποτε ήταν... And, uh, well, I expressed my joy about the re-election of President Obama, but... Ήταν πικρή εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω εύκολα πως η μόνη πρόταση που είπε για την Ευρώπη στην τελευταία του ομιλία ήταν η εξής. Κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω εύκολα πως η κρίση στην Ευρώπη πρέπει να περιοριστεί τελεία. Βεβαίω έχει δίκιο. Οπότε νομίζω πως υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ πέρα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη σοβαρότητα όλων όσων μας είπατε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια και αυτά τα οποία λέει η κυρία Κλίντον, αλλά δεν ξέρω αν το αμερικανικό κοινό γνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ μα. Τι μπορεί να γίνει, λοιπόν? μπορεί να γίνει κάτι για να βελτιωθεί αυτό. Σα ευχαριστούμε κυρία Νίτς. Για τους πράσινους ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρέσβη, θέλω να συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να οικοδομήσετε την ε, διατλαντική σχέση και εξετάζοντας τη δουλειά που έχει γίνει, πράγματι το επιβεβαιώσατε. Αναφέρατε το όραμα του Πρόεδρου Ομπάμα για το μέλλον της εταιρικής σχέσης. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν άκουσα πολλά τέτοια πράγματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Οπότε αναμένω να μας πείτε κάποια περισσότερα. Και ίσως η οικονομική και εμπορική σχέση και πιθανώς μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα μπορούσε να επιβεβαιώσει αυτή τη φιλοδοξία για βελτίωση αυτής της σχέσης. Να αναφέρω σύντομα τέσσερα σημεία Πρώτα απ' όλα εγώ θα ήμουν ε, ευτυχής ε, και οι Ευρωπαίοι φαντάζομαι αν ε, ξαναθυμούνταν τα του κλίματος ο πρόεδρος. Κάπου εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Μια πιο φιλόδοξη διπλωματία από τις είπα θα βοηθούσε τον κόσμο. Το κοινοβούλιο αυτό έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να στηρίξει ε, μια αναβάθμιση του Παλαιστινιακού καθιστώτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και οπωσδήποτε θα θέλαμε να επενεξετάσουν οι ΙΠΑ τη θέση τους. Ε, βλέπουμε εδώ πέρα επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Και τέλος, μια ερώτηση. Η πρώτη θητεία του Πρόεδρου Ομπάμα ξεκίνησε με τη φιλοδοξία του να πατήσει το κουμπί Reset στις σχέσεις με τη Ρωσία. Ε, κάπου δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Η Γερμανίδα καγκελάριο το ίδιο έκανε και γίνεται πιο σκληρή με τη Ρωσία από ό,τι στο παρελθόν. Τι να περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκα από την ομάδα των Κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζουμε. Ε, μιλήσατε για την ψηφοφορία για το SWIFT και εγώ πάντα λέω πως αυτό ήταν ένα καμπανάκι για τις ΗΠΑ αναγνώρισαν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη Λισαβόνα στον τομέα εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής και το ενδιαφέρον της κυβέρνησής σας έχει αυξηθεί έκτοτε. Είχαμε και την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν που μίλησε στην Ολομέλεια. Η ομάδα μου, όπως ξέρετε, έχει ατλαντικό προσανατολισμό. Παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στη δεύτερη θητεία του Πρόεδρου Ομπάμα και ιδιαίτερα ποιο αντικαταστεί στην Υπουργό Εξωτερικών. Νομίζω πως ήταν εξαιρετική Υπουργό Εξωτερικών και προετοιμάζεται τώρα για την να είναι ίσως υποψήφια για πρόεδρος. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα για την δέσμευση της κυβέρνησής σας για ενίσχυση της ειρνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Εμείς συμφωνήσαμε με την θέση της κυβέρνησής σας την προηγούμενη εβδομάδα πως είναι πρόωρο να μιλάμε για αναβάθμιση του καθεστώτος των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ καθώς μπορεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικέ διαδικασίε. Έχω πολλέ ιδιότητε, είμαι και πρόεδρο τη ομάδα φιλία με την Ταϊβάν και ανησυχώ ιδιαίτερα για τι εντάσει στην Ανατολική θάλασσα τη Κίνα και γνωρίζω πω το ίδιο κάνει και η κυβέρνησή σα. Υπάρχουν πολλοί τομεί ε, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Επίση, είμαι εισηγητή για το κέρα τη Αφρική. Μόλι ψηφίστηκε η έκθεσή μου. Πάλι ένα ρόλο, ένας μια περιοχή όπου ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΠΑ ε, και ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικός και απαραίτητος για την καταπολέμηση της πειρατείας, της τρομοκρατίας ε, και πάλι βεβαίως ο ρόλος εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικός τον ΙΠΑ για τη Δυτική Σαχάρα και το Σαχέλ χάρηκα που αναφέρατε τα προβλήματα του Μαλή που θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε και θα απασχολήσει και την κυβέρνησή σας. Αλλά υπάρχουν ε, τόσοι πολλοί τομεί κοινών συμφερόντων, Λατινική Αμερική, η Συμφωνία Ελευθερία με την Κολομβία πρέπει να κυρώσουμε, μέχρι την Νότια Ασία, τις κυρώσει κατά του Ιράν και τη Συρία. Αλλά η ερώτησή μου είναι ο δημοσιονομικός γκρεμό. Τι θα γίνει. Είναι δυνατόν να έχουμε μία ζώνη ελευθερία εμπορίου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν το όνειρο για εμάς τους Ατλαντιστές. Ευχαριστώ. Θα να δώσω τον λόγο στον ε, κύριο Πρέσβη να απαντήσει στις πέντε πρώτες ερωτήσεις και μετά θα ακούσουμε άλλες πέντε ερωτήσεις κύριε Πρέσβη. Οπότε θα έχετε και την ευκαιρία στο τέλος να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα καλά σας λόγια, τα συγχαρητήρια για την εκλογή του Προέδρου μας, το εκτιμούμε αυτό πολύ. Όπως ε, ξέρετε, θα ήθελα να καταλάβετε και να εκτιμήσετε ότι στο συντονισμό μας με το Κοινοβούλιο εκτιμούμε το γεγονός ότι πολλοί από εσάς ασχολείστε με θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας. Ε, όπως η Μέση Ανατολή, ο κ. Σαλαφράγκα ήταν στην Μέση Ανατολή με την κάθε άστον και η κυρία Γκόμες τακτικά επισκέπτεται την περιοχή. Εμείς ε, εκμεταλλευόμαστε πολλές από τις πληροφορίες που μας δίνετε όταν κάνετε αυτές τις επισκέψεις και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω. Αλλά επίσης ανακαλύψαμε πως έχετε σχέσεις με κάποιες από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της ε, Μέσης Ανατολής που εμεί δεν τι έχουμε μέσω των επαφών των πολιτικών ομάδων κτλ. Μα βοηθά πραγματικά λοιπόν όταν επισκέπτεστε αυτέ τι περιοχέ αυτέ και μα ενημερώνετε μετά και μας ε, φωτίζετε. Ε, θα είμαι σύντομο τώρα στις απαντήσεις σας. Κύριε Σαλαφράγκα με ρωτήσατε για την Κούβα και τις πιθανότητες περισσότερης ευελιξίας για το δεύτερο, τη δεύτερη θητεία. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ε, κατά πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση στην Κούβα ε, που, έτσι ώστε να υπάρξει και αλλαγή από δικές μας πλευράς. Ε, σημαντική <coughs> καταστολή στην Κούβα και καταπίεση των αντιφρονούντων, των καλλιτεχνών και άλλων. Μέχρι ότου δούμε λοιπόν κάποια προθυμία για αλλαγή στο επίπεδο της ε, καταπίεσης εκεί, δεν φαντάζομαι ότι θα δούμε κάποιες ε, σημαντικές αλλαγές. Ελπίζουμε ωστόσο ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την πολιτική μας προς την Ασία και την ε, Νότια Κίνα και την θα προσπαθήσω να συνοψίσω την απάντησή μου. Όταν ο πρόεδρος είπε ότι θα εστιάσουμε την εξωτερική μας πολιτική στην Ασία, εγώ είχα να, ε, κάποιες ανησυχίες εδώ να αντιμετωπίσω, ότι δηλαδή ίσως αυτό θεωρούσε πως ε, θα εγκαταλείπαμε ας πούμε την Ευρώπη. Αυτό έχει αλλάξει νομίζω. Υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη αναγνώριση πως η ΕΠΑ όχι μόνο πρέπει να μετακινηθούν προς την, προς την Ασία, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να μετακινηθεί προς την Ασία και έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την Κάθη Άστον. Ε, έχουμε μια κοινή δήλωση στην ΠΝΟΜΠΕ κάνει τον Ιούλιο που δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε για την πολιτική μας για την, απέναντι στην Ασία. Δεν βλέπουμε και η κυρία Γκόμες νομίζω αναφέρατε και χρησιμοποιήσατε τη, τη, τη φράση στρατιωτική απειλή από την Κίνα. Εμείς δεν το βλέπουμε. Ναι, στρατιωτική ε, προετοιμασία. Εμείς φυσικά διατηρούμε μαζί με την Ένωση το εμπάργο όπλων στην, για την Κίνα, αλλά γνωρίζουμε ωστόσο πως η Κίνα είναι μια αναδυόμενη δύναμη με, αυξανόμενη, με, με αναπτυσσόμενη και δυναμική οικονομία και η βασική μας ε, στάση είναι να καλωσορίσουμε την Κίνα ως εταίρο μας μαζί μας και με την Ευρώπη στην αρχιτεκτονική παγκόσμια διακυβέρνηση που πιστεύουμε ότι λειτουργεί για τον κόσμο μέσω διεθνών οργανισμών όπως ε, η ΟΗΕ και, το, ναι. και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κτλ. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε εμπορική εταιρική σχέση με την Κίνα και η συνεργασία μας με την Ευρώπη μπορεί αυτό να το προωθήσει κατά γνώμη μας. Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις ε, ε, όσον αφορά την Ευρώπη και τις εκλογές Όπω είπε και ο κύριος Μπουτικόφερ. Καταρχήν, ε, όπως όλοι γνωρίζετε, οι προεδρικές μας εκλογές δεν είχαν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, αλλά είχαν να κάνουν με την εσωτερική μας οικονομία. Και δεν είναι εντυπωσιακό ότι δεν έγινε πολλή λόγος για την ε, Ευρώπη, για την εξωτερική πολιτική εν γέννη. Γι' αυτό και με εντυπωσιάζει όταν ακούω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί δεν συζητήθηκε περισσότερο η Ευρώπη στις προεδρικές εκλογές. Εγώ ζώντας εδώ έχω παρατηρήσει πολλές εκλογές στην Ευρώπη και η ΕΠΑ δεν συζητώνται στις δικές σας εκλογές. Γιατί περιμένετε λοιπόν εμείς να μιλάμε για την Ευρώπη στις δικές μας εκλογές. Οι εκλογές ε, ε, με αφορούν χώρια, εσωτερικά θέματα. Δηλαδή φόροι, συντάξεις, κοινωνική πρόνοια, αυτά απασχολούν τον κόσμο. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω σχετικά είναι ότι θέματα που φτάνουν να απασχολούν ε, τα θέματα της, της Προεδρίας είναι τα θέματα που, που υπάρχει κρίση. Μα με την Ευρώπη δεν έχουμε κρίση. Η κρίση που μας απασχολεί είναι η οικονομική κρίση όπως και εσάς. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανέφερε την κρίση της Ευρωζώνης και ε, δουλεύει για την κρίση αυτή στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας. Ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μπουτικόφερ για τις κλιματικές αλλαγές που είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Ο πρόεδρος, μάλλον η προεδρική εκστρατεία για την πρώτη θητεία υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμήσει τις κλιματικές αλλαγές. Φαντάζομαι όλοι το γνωρίζετε αυτό. Απογοητευθήκαμε, όπως και πολλοί εδώ, που δεν μπορέσαμε να Πάμε στην Κοπενχάγη, στην COP15, περνώντας, αφού μάλλον είχαμε περάσει και νομοθεσία στη ΣΥΠΑ. Όσον αφορά την εμπορία εκπομπών. Όμως ο Πρόεδρος έχει κάνει πολλά παρόλα αυτά και όσα μπορεί χωρίς να κοντράρεται με το Κογκρέσο για τις κλιματικές αλλαγές πιστεύουμε πως η μείωση των εκπομπών μας ε, βασιζόμενη στο ορόσημα του 2005 έχουν επιτευχθεί και μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Ε, κάτι ακόμα ήθελα να πω για την ερώτηση του κ. Τάνοκ για το φορολογικό ήφαλο, Ναι, εδώ ε, πρόκειται για εσωτερική πολιτική. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Συμβαίνουν διάφορα καθώς μιλάμε γιατί υπάρχει ένα θέμα αναπροσαρμογής στο Κογκρέσο. Ο πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τζον Μπέιν και άλλους για να προσπαθήσει να το λύσει. Ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να αποφύγουμε ένα φοβερό οικονομικό αποτέλεσμα, όχι μόνο για τη ΣΥΠΑ αλλά και για την Ευρώπη. Ίσως αυτά μόνο να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Έχουμε ακόμα πέντε συναδέλφους και θα ήθελα να ρωτήσω, να του ζητήσω να διατηρήσουν τις παρεμβάσεις τους στο ένα λεπτό. Γιατί έχουμε και μια συνάντηση με τον, με τον Υπουργό της Μακεδονίας. Ο κ. Μιλανμόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Μιλιάς. Είναι πολύ σημαντικό το πόσο βαρύ είναι η σχέση μας και για σας. Και όπως είπε ο κ. Κλίντον, είναι η απαραίτητη δύναμη η Ευρώπη και ε, να δούμε τώρα ακριβώ τι θα γίνει όσο την εξυγίανση των δημοσιονομικών και ποιε θα είναι οι συνέπειε για την ε, εξωτερική πολιτική. Με είπατε μέσα τι, τι γίνεται με τις άλλες επίρρους, τα το θέματα που υπάρχουν και κυρίως για την Κούμα. Για πέστε μας, ε, σε αυτή την δεύτερη θητεία, η κυβέρνηση Ομπάμα, πώς, πώς βλέπει τη σχέση με την Λατινική Αμερική. Ευχαριστούμε πολύ κύριε για σα, Ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο σύντομο, κύριε Κύριλοφ. Το πολύ ένα λεπτό, κύριε Πρεσβή. Και εγώ σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και θέλω να σα πω σε σχέση με ε, αυτά τα οποία πάρα πολύ εύστοχα μα είπατε όσον αφορά την αλλαγή τη αιστεία τη προσοχή τη πολιτική μα. Για πετε μα, είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι ο ίδιο ο πρόεδρο Ομπάμα να έρθει σε Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες κατά αυτή τη δεύτερη θητεία και έτσι ακριβώ να αποδείξει το πώ σημασία αποδίδει στη σχέση μα. Επίση, σα ευχαριστούμε για όσα εξηγήσατε, αλλά υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, θέλω να σα ρωτήσω. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα, χρειάζονται οι κάτοικοι του θεωρεί διαβατηρίων για να ταξιδέψουν στη ΣΥΠΑ. Γίνεται κατά τη δεύτερη αυτή θητεία να πετύχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το, το μέτωπο, γιατί αυτό είναι ένα αναχρονισμό. Ε, εντάξει, είναι το θέμα του, του, του πόσες είναι οι, οι αιτήσει που, που απορρίπτονται, αλλά τελικά οι, οι σα σας υπρόξενο κανείς. Έχετε εσεί και το μαχαίρι και το πεπόνι, όπως λέμε. Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια ε, κύριε Πρέσβη, συγχαρητήρια για την εκλογή του Πρόεδρου και βεβαίω ε, είναι πάρα πολύ σημαντική συνέπεια ότι εσείς θα συνεχίσετε να είστε εδώ όσο συνεχίζει να είναι πρόεδρος ο κύριος Ομπάμα. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αυτή την οποία ε, ρώτησε και ο κύριος ε, Κύριλοφ. Καλέσαμε όταν είμαστε, ήμουν πρόεδρος τον κύριο ε, τον πρόεδρο που να έρθει δεν μπορούσε να έρθει είχε έρθει ο Κλίντον αλλά όχι, όχι το, το, το, ούτε ο πρόεδρος Κλίντον το 95 είναι ο τελευταίος πρόεδρος που ήρθε ο πρόεδρος Ρίγκαν στο Στρασβούργο οπότε έχουν περάσει 30 χρόνια και θα είναι πολύ καλό να έρθει ξανά ο πρόεδρος ε, να μα μιλήσει. Κύριε, πολύ ευχαριστώ ότι ο πρόεδρο Σούλτ ε, θα συναντήσει τον κύριο Ομπάμα, τον πρόεδρο Ομπάμα σήμερα. Συγχαρητήρια επίση γιατί κάνετε στην ε, Μέση Ανατολή. Για πετε μα, ποια είναι η θέση των ΗΠΑ όσον αφορά την Χαμά. Δεν αποτελεί αντίφαση το ότι από τη μια μεριά λέτε ότι θέλουμε λύση που να περιλαμβάνει και τα δύο κράτη, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουμε να προσδώσουμε ένα καλύτερο καθεστώ στους ε, Παλαιστινίους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να περιλάβουμε περισσότερο τους Παλαιστινίους στην διαδικασία. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε θα είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τόσα ενθαρρυντικά μας είπατε. Ευχαριστούμε κύριε Πέτρη, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σχάκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και εγώ να σας συγχαρώ για σας ε, και την κυβέρνησή σα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ψηφιακή ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Μήπω μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Και τελικά να μην κατησχίσει τη ελευθερία η κυβερνοασφάλεια, γιατί υπάρχουν τέτοιε παρεξηγήσεις. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τον διάλογο των ε, νομοθετών τον διατλαντικό. Έχουμε μια εκδήλωση αυτή τη βδομάδα, να δούμε πώ θα βελτιωθεί η συνεργασία. Ε, να δούμε πώς δεν θα αποσπάτει η προσοχή μας προς άλλες κατευθύνσεις ε, γιατί τα πρώτα γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Κατά τη συνεργασία μας θα πρέπει να είμαστε και ανεξάρτητοι του άλλου αλλά και συμπληρωματικοί. Νομίζω καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί ε, και η κυβέρνηση και το Κογκρέσο ότι υπάρχουν ε, αντίκτυποι όσον αφορά το, τις κυρώσεις που επιβάλλουμε ε, στο Ιράν ή γενικά στις ισχυρώσεις για, για την πνευματική ιδιοκτησία. Και εμείς ε, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά θέλουμε να μην λαμβάνονται μέτρα τα οποία είναι βλαπτικά και για εμάς και για εσάς. Πώς επομένως θα ενεργήσουμε τέτοιο τρόπο, ώστε οι κοινοί στόχοι να εξυπηρετούνται. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λούνατσεκ, σας ευχαριστώ και ο πλευρά των Πρασίνων, καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια για όλα όσα μα είπα. Συγχαρητήρια και για την εκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα. Δύο θέματα θα σας αναφέρω. Το ένα το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Το θέμα του τι θα γίνει την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπατε, ε, είχατε ένα ψήφισμα ε, είχαμε εμείς μόνο εδώ ένα ψηφνό και υπήρξε ε, ευρεία υποστήριξη και θέλουμε να αποκτήσει η Παλαιστίνη το καθεστώς του παρατηρητού. Εγώ είμαι τώρα το άλλο θέμα, η συγγήτρια για το Κόσοβο. Ε, εκτιμώ το ρόλο των ΙΠΑ στο Κόσοβο και επίσης ε, έχει έρθει στην διάσκεψη που έγινε η Μαντίν Ολμπράιτ η κυρία Κλίντον, η Λέδη Άστον, ε, όλοι είχαμε κοινή προσέγγιση. Και από τα θεσμικό όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει περισσότερο από όλους την ανεξαρτησία. Όμως υπάρχουν πέντε χώρες που δεν συμφωνούν ε, για την ανεξαρτησία της χώρας. Εσείς τι λέτε, θα αποκτήσει ποτέ το, το καθεστώς του αναγνώρισε αναγνώρισης ως ανεξαρτήτου χώρα στο Κόσοβο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Πρόεδρος θα έχει ευκαιρία να σας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μιλαν Μιλανμόν ρώτησε για τον νομοσυνομικό γκρεμό. Θα το συνοψίσω. Είναι κάτι αρνητικό εάν συμβεί γιατί κατά βάση όπως θυμάστε τον Αύγουστο πέρσι τον Αύγουστο είχαμε πρόβλημα με την οροφή του χρέους το Κογκρέσο και ο Λευκός Σύκος αποφάσισαν να αναβάλουν το ζήτημα μέχρι φέτος. Εάν το Κογκρέσο δεν δράσει, τότε θα έχουμε αυτόματες περικοπές και αυξήσεις φόρων. Συνολικά Μιλάμε για ένα πλήγμα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομία που θα μπορούσε να ξαναρίξει τη χώρα στην ύφεση, σύμφωνα με κάποιους. Γι' αυτό υπάρχει κίνητρο για να λυθεί αυτό το ζήτημα. μετεκλογικά για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση που θα είναι δυσάρεστη και για μας και για την Ευρώπη. Για τη Λατινική Αμερική πρέπει να ομολογήσω κάτι. Πέρασα τον χρόνο που προσπαθούσα να καταλάβω την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη και δεν έχω εστιάσει τόσο πολύ στη Λατινική Αμερική. Όμως ε, μπορώ να σας φέρω σε επαφή με του ειδικούς μας, αν θέλετε. κύριοι Κύριλοφ και Πέτερινγκ ζήτησαν να μάθουν εάν ο πρόεδρος θα, επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο στη δεύτερη θητεία του. Εγώ θα το ήθελα περισσότερο από όλους ε, τους παριστάμενους στην αίθουσα. Και ελπίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε κάποια στιγμή, αλλά επειδή το πρόγραμμα του Προέδρου είναι αυτό που είναι, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Είναι απρόβλεπτο. Ελπίζω όμως να συμβεί. Προσπαθώ. ρωτήσατε για το καθεστώ βίζας, αντιλαμβάνομαι την απογοητευσή σας. Ο πρόεδρος το αντιλαμβάνεται. Ε, στην πρώτη θεία προσπάθησε να απελευθερώσει το καθεστώ αυτό σε σχέση με την Πολωνία. Αντιλαμβανόμαστε την απογοητευσή σας. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στην ομοθεσία μας Γιατί το κάνουμε αυτό, προστατεύουμε τα σύνορά μας και κάθε κυρίαρχο κράτο ε, το ίδιο κάνει, αποφασίζει ποιο μπαίνει έντο της χώρας. Και θα συνεχίσουμε να το κρίνουμε εμείς. Έγιναν κάποιε ερωτήσει. για το Παλαιστινιακό και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προφανώς είναι δύσκολο το ζήτημα για εμάς. Γιατί ερχόμαστε σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια κρατημέλη, αλλά έχουμε αποφασίσει πως ε, μόνο λογική και παραγωγική οδός για ειρήνη είναι άμεση συνομιλίες Παλαιστινίων Ισραηλινών. Θεωρούμε πως η αναγνώριση ε, από τον ΟΗΕ δεν θα αλλάξει ουσιαστικά το γεγονός πως πρέπει δύο πλευρές ε, να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε μια ειρήνη. Επίση θα υπάρξουν και κάποιε συνέπειε για τη χρηματοδότηση τη Παλαιστινιακή αρχή, Οπότε θεωρούμε πω το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρεθούν ξανά μαζί σε ένα τραπέζι δύο πλευρέ και να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά μαζί. Θα απαντήσω στο ερώτημα τώρα για την Σερβία Κοσφοπέδη και μετά θα επανέλθω στο άλλο για την ψηφιακή ελευθερία. Και εμείς ικανοποιηθήκαμε από τη συνεργασία μας για τα στα δύσκολα ζητήματα Σερβίας Κοσφοπεδίου αλλά αναγνωρίζουμε επίσης πως εσείς έχετε βεβαίως ε, το μοχλό πίεσης που λέγεται ένταξη. Αλλά και οι δύο χώρες πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και ελπίζουμε να γίνουν μέλη της ε, διεθνικής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 90 χώρες που αναγνωρίζουν το κοσφοπέδιο ε, και ελπίζουμε πως ε, εάν ομαλοποιηθούν σχέσεις με τη Σερβία θα επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης από τις άλλες χώρες και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Τέλος, για το ε, ερώτημα της κυρίας Χάκη για την ψηφιακή ελευθερία. Μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Εμένα απασχολεί δεδομένου του ότι σε μια προηγούμενη ζωή μου στον κόσμο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να πω πως τον επόμενο μήνα η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση θα συνεδριάσει στο Ντουμπάι και θα εξετάσει τα ζητήματα δηλαδή, του πώς πρέπει να κυβερνηθεί το διαδίκτυο και εμεί θεωρούμε πως ο καλύτερος τρόπος για να κυβερνηθεί το διαδίκτυο και να προωθηθεί η ψηφιακή ελευθερία είναι να συνεχιστεί το σύστημα το οποίο το έχει κάνει τόσο επιτυχές μέχρι στιγμής. Δηλαδή ενίσχυση της διαδικασίας πολλών συμμετεχόντων και λιγότερη εποπτεία από τα κράτη. Χαιρόμαστε για το ψήφισμα που υιοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο που ενίσχυσε την ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για κυβέρνηση του ίντερνετ είναι μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μηχανικών, κοινωνία των πολιτών και ανθρώπων που έχουν ε, κάποιο συμφέρον και όχι μέσω ελέγχου από τα κράτη. Έτσι θα ενισχυθεί η ελευθερία του διαδικτύου. Ξέρω πως δεν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, αν θέλετε να συζητήσουμε κάποια στιγμή με μένα ή σε κάποια εβδομάδα μου, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας μιλήσω σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη που ήρθατε εδώ σήμερα και βέβαια αναμένουμε τη συνέχεια της συνεργασίας, συνεργασίας μας. Συνάδελφοι, σε σύνδεση με την αντιπροσωπεία της κοινή κοινοβουλευτική επιτροπής με την ΦΥΡΟΜ έχουμε σήμερα μαζί μας τον Νικόλα Προπόσχη, Υπουργό Εξωτερικών της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και θα μιλήσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα και για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια να σας ε, καλωσορίσω, Υπουργέ και καθώς και τον κύριο Μαρκάκη, που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας στην κοινή κοινοβουλευτική, μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου και ε, Φύρομ. Θα ήθελα να τονίσω πως η διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μας ε, οδηγήσουν στο ότι διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία. Επίσης στηρίζουμε μία κοινή αποδεκτή λύση για το θέμα του ονομασίας με την Ελλάδα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω και να υπογραμμίσω πως η πρώην ε, Δημοκρατία της Ιουκοσλαβίας Μακεδονία ε, σκοπεύει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις ε, για να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει αποτελεσματικό και ανεξάρτητο δικαστικό σώμα που θα καταπολεμήσει την διαφθορά, θα ε, ε, καταπολεμήσει την πολιτική επιρροή στα ΜΜΕ και η ενταξιακή πορεία είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Επίσης θέλουμε να παραμείνει ψηλά η προοπτική της ε, ένταξης και να παραμείνει η χώρα δεσμευμένη στην ενταξιακή διαδικασία. Και δίνω το λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών που πώς για μια σύντομη παρουσίαση και έπειτα θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι για ερώτα σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ε, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω την κατάσταση στη Μακεδονία τον τελευταίο χρόνο και να σας δώσω επιχειρήματα γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε στην διαδικασία ε, Εκτιμούμε τις δηλώσεις και τις θέσεις που έχετε κάνει και αντικατοπτρίζουν ήδη τις θέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα είμαστε δύο εβδομάδες πριν από το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πρέπει να λάβει απόφαση για τη διαδικασία διεύρυνσης και διάφορα θέματα είναι επιτάπητος, εύκολα και λιγότερο εύκολα. Εγώ θα την να πω η διαδικασία διεύρυνσης δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, αλλά ήταν η πιο επιτυχής από όσε έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν. Ο στόχο αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων θα είναι να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με τη Μακεδονία. Θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, πω μετά από 7 χρόνια ω υποψήφια χώρα είμαστε πια έτοιμοι να αρχίσουμε τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αυτό χρειάζεται. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, το 2012 ήταν δυναμικό και ε, έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές, έχουμε φτιάξει μια μεγάλη ατζέντα για μεταρρυθμίσεις και έχουμε δεσμευθεί για τις ε, σχέσεις καλής γετνίασης. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε πως η Μακεδονία εξακολουθεί να πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια και σύστησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Υπάρχει μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις προηγούμενες συστάσεις που είχαν γίνει. Εγώ σύντομα να τονίσω τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε το, σημαντική τομή. Η αποτελεσματικότητα του δικαστικού σώματος έχει βελτιωθεί. Ε, οι καθυστερημένες υποθέσεις μειώθηκαν κατά 12% και κατά 35% στις πιο σημαντικές υποθέσεις. Έχουμε επίσης τροποποιήσει την νομοθεσία μας όσον αφορά τον ορικαθορισμό προθεσμιών για κάθε μια από τις διαδικαστικές φάσεις που θα επιτρέψουν στο δικαστικό δικαστικό μας σύστημα να διεκπαιρεώσουν όλες τις καθυστερήσεις. Έχουμε τονίσει λοιπόν τον επαγγελματισμό του δικαστικού σώματο. Αυτό έγινε μέσω των αποφύτων της Ακαδημίας για την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων που σταδιακά σωματώνονται στο δικαστικό σύστημα και από του χρόνου οι δικαστές και οι εισαγγελείς μπορούν να προσληφθούν μόνο ως οι απόφοιτοι αυτής της σχολής. Για να ενισχύσουμε την ελευθερία έκφραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε ποινικοποιήσει την δυσφήμιση και την προσβολή λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εννοείται πως αυτό έχει συνδυαστεί με διάφορες ε, καταρτήσεις ε, του δικαστικού, κυρίως ε, δικαστές και προσπαθήσαμε όχι μόνο να θεσπίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά δικαστικά στάνταρ αλλά και να εξασφαλίσουμε πώς θα τηρηθούν αυτά. Στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της... Έχουμε μιλήσει για Μάλλον έχουμε αυξήσει την διαφάνεια αυτού του σημαντικού εργαλείου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η πρώτη έκθεση για την δεκαετία της ε, εφαρμογής της ε, Συμφωνίας Πλαισίου της Οχρίδας έχει γίνει. Η αρχή Επίσης, τη μη διάκριση ε, στις ε, διοικήσεις ε, έχει εφαρμοστεί, έχει δοθεί έμφαση στις μικρότερες εθνοτικές κοινότητες. Σημαντικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει. Νέος κανόνας νόμος για την διοίκηση έχει ήδη συνταχθεί για να παγιωθεί και να εδραιωθεί ο προεπαγγελματισμό στη δημόσια διοίκηση. Επίσης, έχει βελτιωθεί η αξιοκρατία στην δημόσια διοίκηση και ο σεβασμό τη αρχή τη ισότιμη εκπροσώπηση. Σε σχέση με τι εκλογικέ μεταρρυθμίσει. έχουμε τροποποιήσει τον εκλογικό νόμο και τον νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Κάτι που είναι περίπλοκο σε όλε τι δημοκρατίε. Έχει αυτό αντιμετωπιστεί σωστά και έχουμε λάβει υπόψη όλε τι συστάσει από την ΟΑΣΕ. Και επίσης έχουμε καταγράψει όλες αυτές τις διατάξεις ε, το... Ε, θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την οικονομία αγοράς. Έχουμε λάβει μέτρα για βελτίωση της αγοράς εργασίας, να μειώσουμε την ανεργία και να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό μας περιβάλλον εστιασμός μας έμφαση δίνεται στην λάπνεση της παγκόσμιας κρίσης. Όπως ξέρετε είμαστε 90% συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπόριό μας γίνεται με τις χώρες ευρωπαϊκές και τις υποψήφιες χώρες και γι' αυτό και έχουμε άμεσες επιπτώσεις από την κρίση. Όπως εσείς γνωρίζετε, η απουσία ενταξιακών διαπραγματεύσεων το Μάρτιο ξεκινήσαμε έναν υψηλό επίπεδο διάλογο με την Κομισιόν. Έχουμε πολύ στενές πλέον επαφές και ε, έχει δοθεί έτσι η όθηση στις μεταρρυθμίσεις. Είχαμε τρεις διαλόγους με την συμμετοχή του Επιτρόπου Φίλες στα Σκόπια. Ωστόσο αυτός ο διάλογος θα πρέπει να τονίσω πως είναι εξαιρετικά χρήσιμο μέσο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πραγματικές ε, ενταξιακές διαδικασίες για μια υποψήφια χώρα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε αυτά αποτελέσματα, να πληρώσουμε δηλαδή ε, τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης και να ανταποκριθούμε στις συστάσεις της Κομισιόν. Η κυβέρνηση της Μακεδονίας πρόσφατα υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράσης, αλλά Ελπίζουμε πως έτσι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην ε, έναρξη της διαδικασίας ένταξης. Έχουμε τώρα πρόβλημα και, με τους, ε, και ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε και τις σχέσεις μας με τους γειτονές μας. Είμαστε στην καρδιά των Βαλκανίων και γι' αυτό και θα πρέπει να αναπτύξουμε τις πολυεθνικές μας κοινωνίες που αντικατοπτρίζουν τους πολιτιστικές μας συνδέσμους με τους γειτονές μας. Θέλουμε εταιρικές σχέσεις με τους, με τους γειτονές μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε στους δύσκολους αυτούς αυτούς καιρούς διμερώς, περιφερειακά, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για κοινή ευημερία. Έχουμε ήδη συμβάλει πολύ και, προσπαθ... και να το πράξουμε και στο μέλλον. Έχουμε λύσει όλα τα συνοριακά θέματα. Έχουμε επιτύχει πλήρη συνοριακή χάραξη. Μπορεί να το... σας ακούγεται μυστήριο αυτό, αλλά στα Βαλκάνια αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και σπάνιο. Έχουμε συμβάλει λοιπόν στις αποστολές ασφαλείας στην περιοχή. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην οικοδόμηση των, της κατασκευή μάλλον των πανευρωπαϊκών ε, διαδρόμων ε, βορρά, νότου και ανατολής δύσης και θέλουμε να έχουμε ανοιχτά σύνορα με τους συναδέλφους. Σε σχέση μας με τώρα με την Ελλάδα θα είμαι σαφής επιθυμία μας είναι να προχωρήσουμε μαζί με την Ελλάδα στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υποβάλει διάφορες προτάσεις για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και οικοδόμηση κλίματος αμοιβαία εμπιστοσύνης. Έχουμε ανταποκριθεί θετικά στην πρόσφατη ελληνική πρόταση για ένα memorandum κατανόησης για να προχωρήσουν οι συζητήσεις για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία του ονόματος. Παραμένουμε με καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις ε, της διαμεσολάβησης του ΟΗΕ και είμαστε προσιλωμένοι στην εξέβρεση μιας ε, λύσης σε σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και του διεθνούς νομικού πλαισίου που ορίζεται από το Ηνωμένο ε, Εθνών. Τις διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Θα είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Επίση, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σχέση μα με τη Βουλγαρία. Υπάρχουν θέματα κοινού συμφέροντο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πιστεύω πω θα πρέπει να αφήσουμε την ιστορία πίσω μα και στου ιστορικού και ε, πιστεύω πω ήδη έχουμε ένα πολύ καλό νομικό πλαίσιο για να απτύξουμε τη σχέση μα και να ε, επιδιώξουμε κοινά προγράμματα ώστε να ωφελήσουμε του λαού μα. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι για συνεργασία και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο μήνυμα στου Βούλγαρου φίλου μα και όλου όσου υποστηρίζουν την ιδέα της διεύρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνία των πολιτών έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού. Για να, το μήνυμα για να ανοίξουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις θα είναι το πρώτο καλό μήνυμα για τη Μακεδονία αφού έγινε η Βουλγαρία μέλος. Ελπίζουμε, αναμένουμε ότι ως καλός γείτονας και ως μια χώρα που θέλουμε εμείς να έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το, τον θετικό ρόλο που έχει παίξει η Μακεδονία στην τοπική περιφερειακή συνεργασία για την διαδικασία της ε, νοτιοανατολική περιφέρεια τη Ευρώπη είναι η παλαιότερη διαδικασία συνεργασία. Ο ε, βασικός μας είναι να πετύχουμε όλες οι χώρες που δεν έχουν μπει στην συνεργασία να ε, προσχωρήσουν σε αυτήν. Αυτό θα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία και νομίζω πως μια ασφαλής και ευημερής ε, Ευρώπη εξασφαλίζεται από ασφαλή και ευημερή Βαλκάνια. Και αυτό είναι ένας στόχος που είναι κοινό με όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας. Να τονίσω επίσης ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ισχυρή, ένας ισχυρός ενωπητικός παράγοντας η Μακεδονία, δεν έχει την αποκλειστικότητα, είναι εξαιρετικά σημαντικό στην πράξη σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις ε, χώρες που είναι υποψήφιση που επιθυμούν να γίνουν. Πιστεύω όμως πως η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα έχει πολλαπλό θετικό αποτέλεσμα γιατί θα λειτουργήσει ως καταλήτης στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, θα ε, καταστήσει εντονότερες τις δυναμικές μεταρρύθμισης και θα έχει ενωτικό, ε, ενωτική επιρροή όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Ε, περαιτέρω θα αυξήσει την όθηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Βαλκάνια και θα υπογραμμίσει την αξιοπιστία της ε, πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι σίγουρα θα δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στις διμερείς συζητήσεις με την Ελλάδα ώστε να ξεπεραστεί η διαφορά μας για το όνομα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, και, και η ώρα για μια νέα επικοδομητική προσέγγιση και στρατηγική Στρατηγικό προβληματισμό πολλές φορές έχουν ληφθεί αποφάσεις διαχειριστικές. Αλλά τώρα πρέπει να επιστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικό ε, προβληματισμό όταν γίνονται, λαμβάνονται αποφάσεις για τη διεύρυνση. Άλλο είναι να ε, επιβεβαιώσουμε τις εμπειρίες των προηγούμενων κύκλων διεύρυνσης και ότι δηλαδή εν γέννη τα εμπόδια δεν ε, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο να ευνοεί την υπέρβαση των διαφορών και την ε, άβληση των διμερών διαφορών. Το αντίθετο ισχύει. Η διευκόλυνση της εισόδου στην Ένωση το αμβλύνει και, το, και, και, και μάλλον διευκολύνει την επίλυση επίλυση των διμερών σχέσεων και σίγουρα δημιουργεί το κλίμα που χρειαζόμαστε σε αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη. Παράλληλα μπορούμε να επιδιώξουμε και τη λύση των διμερών θεμάτων. Για να είμαι ξεκάθαρος δεν υπάρχει κανείς που να έχει μεγαλύτερο συμφέρον από ότι η ίδια η Μακεδονία για να ξεπεραστούν οι διαφορές για το όνομα που έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στη διαδικασία ολοκλήρωση των παρελθών και νομίζω πως θα ήταν ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί και στην υπόλοιπη περιοχή ότι δεν παίζουμε καθυστέρηση, δεν θέλουμε δηλαδή να καθυστερήσουμε, αλλά τονίζουμε τις πτυχές που είναι πιο σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία και για το κοινό μας μέλλον. Η Μακεδονία δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση παρά να ακολουθήσει το δρόμο προς την ε, Ένωση. Και το δρόμος αυτό στα τελευταία 20 χρόνια ε, έχει στρωθεί, είναι ένας δρόμος που έχει ισχυρή στήριξη από όλες τις χώρες, γιατί, ε, από όλη τη χώρα μας, γιατί 90% του πληθυσμού μας στηρίζει την ένταξη στην Ένωση. Και νομίζω πως φέτος η εξολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάνει μια ανανεωμένη έκκληση πια ε, λέγοντα όλα τα κρατημέλη πω οι διαπραγματεύσει ενταξιακέ θα πρέπει να ξεκινήσουν και να πούμε πω τα ωφέλη θα ωφελήσουν όλα τα κρατημέλη γιατί θα ωφελήσουν ε, και ταυτόχρονα και του ε, πολίτε τη Μακεδονία. Ορισμένοι μπορεί να ισχυρίζονται πω δεν είναι κατάλληλη στιγμή για τη διεύρυνση. Τα ακούω αυτά σε, σε, σε, επίσημα και άτυπα βήματα, αλλά Είμαστε μέρος τη εσωτερική αγορά, οτό ή άλλου. Ε, Στανόμαστε και νιώθουμε τι αισθανόμαστε και νιώθουμε τις ε, επιπτώσεις της κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Αλλά η καλύτερη τι επιπτωσει τη κρισης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι να συνεχιστεί η καλυτερη επενδυση σε αυτους τους δυσκολου καιρου ειναι να συνεχιστει η διευρυνση με τη Μακεδονία και τι Βαλκανικέ χώρε μέσα στη λέσχη και Όταν κανείς έχει κάνει αυτά που έπρεπε πρέπει και να ανταμειφθεί. Πρόκειται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το, το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη τονίζει την ανάγκη να ολοκληρώσει την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω πως η Μακεδονία μπορεί να παίξει αυτό τον ενωτικό ρόλο. Επίσης είναι πολύ σημαντική πτυχή για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίω, διότι ορισμένοι λένε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα καταφέρει τοπικά στην άμεση γειτονία της, ε, τότε κινδυνεύει και να υποβαθμιστεί ε, παγκοσμίω. Εμείς στα Βαλκάνια πρέπει να προχωρήσουμε στι μεταρρυθμίσεις, αυτό δεν υπάρχει εναλλακτική εκεί, αλλά πιστεύω πως και η Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει πιο πολύ προς την ένταξη με βάση τη μεμονωμένη τις, ε, τα επιτεύγματα μάλλον του καθενός. Και αυτό έχει γίνει και στους προηγούμενους κύκλους και έχει, έχει ένα λογικό θετικό αντίκτυπο επιτόπου. Σίγουρα πρέπει να διατηρηθεί η αξιοπιστία της πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης και φυσικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα μπορέσουν να μετακινήσουν την περιοχή αυτή πιο κοντά στην Ένωση. Εξάλλου θα είναι οι κύριοι ε, ευεργετημένοι μιας τέτοιας διαδικασίας. Η Ελλάδα ως το παλιότερο μέλος ε, στην περιοχή μας θα δώσει, πιστεύω, μια αποφασιστική, καθοριστική βολή όσον αφορά την ανανέωση της ατζέντα 2014 της, της Προεδρίας που είναι προτεραιότητα οι μεταξιακές διαδικασίες. Θα ήθελα να κλείσω παραθέτοντας τον Winston Churchill που είπε ότι το τίμημα της ε, σπουδαιότητος είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία για όσους είναι εκτός της λέσχης αλλά και για όσους είναι εντός της λέσχης. Θέλουμε και είμαστε προσιλωμένοι στη δημιουργία τέτοιου περιβάλλοντος ώστε όλοι να πιστέψουν αυτή τη διαδικασία και είμαστε πεπισμένοι πως ε, κάποια στιγμή από εδώ και μπρος θα επιβεβαιωθεί ότι έχουμε προβεί στις σωστές ε, αποφάσεις έχουμε κοινή ευθύνη, έχουμε και κοινό μέλλον. Και πιστεύω στεναρά πω για να συνεχιστεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ε, θα ωφελήσει αυτό τόσο τους πολίτες της ε, Δημοκρατίας της Μακεδονίας όσο και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα πάψω τώρα και θα ε, δεχτώ ερωτήσεις σας. Σε οποίε ευχαρίστω θα απαντήσω. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και εγώ συμπρόεδρος της ε, μεικτής αντιπροσωπείας θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία κύριε Υπουργέ. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεπαντόφ ε, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ήσασταν πολύ επαγγελματικός και είπατε πώς σε καιρούς οικονομικής κρίσης ε, αντιστέκεστε σε αυτήν. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Αυτό το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι πώς ο λαός ε, σε ποστό πάνω από 90% είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας. Αυτό είναι εξαιρετικό και είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη διάθεση που υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάποια σχέση θα έχει με την πολιτική σας. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Αυτό φαίνεται και στην έκθεσή μας, στις συζητήσεις μας. Είχαμε μια συζήτηση με την Κομισιόν Πάντα βέβαια μας υποδέχεστε με τρόπο φιλικό και θετικό όταν επισκεφτόμαστε τους συναδέλφους μας ε, από την Σομπρανία και βεβαίως ε, ε, σημαντικό είναι ο ενταξιακό διάλογο υψηλού επίπεδου. Λέτε σωστά, κύριε Πρόεδρε, πω δεν είναι υποκατάστατο και δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Αυτό ο διάλογο βεβαίω έχει δημιουργήσει μια δυναμική και αποτελεί ένα κίνητρο θα έλεγα από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και δική σας και βεβαίω θα ήθελα να αναφέρω εδώ πέρα τη δέσμευση της ε, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κυρίας Αρίφη. Βεβαίως υπάρχουν προκλήσεις, ε, πρέπει να τις αναφέρουμε. Να υπόψη την πρόοδο που υπάρχει στα ζητήματα κατσουκιά, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την μεταρρύθμιση της διοίκησης και της δικαιοσύνης, αλλά υπάρχει σαφής πρόοδος, η καταπολέμηση της ε, διαφοράς βεβαίως ε, πρέπει να συνεχθεί, αλλά αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο στη δική σας χώρα στο θέμα ΜΜΕ και ελευθερίας του τύπου πριν από ένα χρόνο ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση το συζητήσαμε αυτό ανοιχτά και ο ανοιχτός αυτός διάλογος οδήγησε σε μια στρογγυλή τράπεζα και εδώ πέρα η αντιπρόεδρος κυβερνήσεως κυρία Ρήφη ενεπλάκη και με χαρά και ανακούφιση διαπιστώσαμε πως οι στρογγυλές αυτές τράπεζες μεταξύ τραπεζών ε, με ε, ΜΜΕ και κυβερνήσεως οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς συνεννοούνται μεταξύ τους οι ομάδες ε, οι ε, Το 2010 λοιπόν σε αυτόν τον τομέα είχαμε αξιοσημείωτα περιστατικά τα οποία μπορεί να ερμηνεύουμε υπερβολικά, αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είχαμε διαδηλώσει ε, βία μεταξύ εθνοτικών, των εθνοτικών ομάδων και το περασμένο Σάββατο είχαμε κάψιμο σημεών. Αυτό είναι πάντα ένα μήνυμα πως ε, η συμφωνία της ε, Αχρίδας ε, και η εφαρμογή της πρέπει να μας απασχολήσει. Να κάνω δύο παρατηρήσεις για τις σχέσεις με τους γείτονες. Ε, βεβαίως το ζήτημα του ονόματος παραμένει εμπόδια. Προσφάτως είχαμε μια κάποια δυναμική μέσω μιας αλληλογραφίας μεταξύ ημών κύριε Υπουργέ και του ομολογούσα στην Αθήνα. Είναι μια σημαντική αρχή αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία τώρα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά τις σχέσεις με τη Βουλγαρία. Εκεί πέρα αλλάζει το κλίμα στην αντιπροσωπεία μας αλλά και εντός της Επιτροπής οι σχέσεις με τη Βουλγαρία ε, φαίνεται πως ε, διαταράσσονται. Και γι' αυτό θα θέλαμε να δώσουμε λίγο βάρος εδώ πέρα και να προσπαθήσουμε ο διάλογος με τη Βουλγαρία να πηγαίνει προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. Προς την κατεύθυνση της περισσότερης ε, ε, Επίσης να αναφερθώ στον Ρίτσαρτ Χάουιτ με τον οποίο πάντα συνεργαζόμαστε εξαιρετικά. Είναι μεγάλος ταξιδιώτης και φίλος της διαδικασίας ένταξης και βεβαίως ε, ε, είναι και σημαντικό συνεργάτη σας και στην αντιπροσωπεία μας. Και πάντα είναι καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο Πρόεδρος. Συνάδελφε. And, uh, I have so many... Έχουμε λιγότερα από 25 λεπτά για τις ερωταπαντήσεις και είναι ένα σωρό που έχουν εγγραφεί να λάβουν το λόγο. Οπότε σα παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κύριος Σαλαβράγκα είναι ο πρώτο που ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κύριε Υπουργέ Ποπόφσκι. Λάβαμε υπόψη προσεκτικά κάθε πρόοδο που έχει κάνει πρόοδο η χώρα σας, ε, δικαιοσύνη, ε, διοίκηση. Ξέρετε εσείς τις θέσεις μας. Γνωρίζουμε καλά τις εκθέσεις που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε το ότι σήμερα πριν μπείτε ε, είχαμε συζήτηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ για την οικονομική κρίση που μαστίζει τον κόσμο, για το πρόβλημα της ε, γάζης, για την διαδικασία ειρήνευσης ε, στην Μέση Ανατολή, Αραβική Άνοιξη, Ιράν κλπ. Οπότε, θέλω να σας πω κάτι. Είναι κάτι μεταξύ ερώτηση και διαπίστωσης. Πώ είναι δυνατόν ενώ η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει με μια τόσο σημαντική πρόκληση σαν τι επαφέ με τη χώρα σε διαπραγματεύσει. δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να, να, να, να, συμφωνήσουμε όσον αφορά την ονομασία ε, μας είπατε καλή θέληση, διάλογος και πάντοτε όταν υπάρχει θέληση βρίσκεται ο δρόμος για να εξευρεθεί λύση και η, η Ελλάδα επίσης μια που είναι μέλος από είναι στην καλύτερη θέση, με καλύτερες διαθέσεις οπότε θα πρέπει τελικά να βρούμε μια οριστική ημερομηνία ούτως ώστε αυτή η διαφορά να επιληθεί που εκκρεμεί τόσο καιρό και αυτό θα ε, είναι προς το συμφέρον ε, όλων στρατηγικό ε, συμφέρον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος ως μέλους κράτους. Οπότε αυτό ήθελα να θέσω επιτάπητος κύριε Υπουργέ γιατί νομίζω ότι θα πρέπει άπαξ και διαπαντός να σταματήσει αυτή η εκκριμότητα η οποία μας ταλανίζει τόσο καιρό. Κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα χαίρομαι να βλέπω τον κύριο Παπόσκη στην Επιτροπή μας, συναντιόμαστε τακτικά και όπως είπε και ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, συναντιέμαι μαζί του με τον κύριο Κρουέσκι, με όλα τα κόμματα και πολλούς ανθρώπους στη χώρα τακτικά και με ικανοποιεί αυτό. Επειδή πρέπει να είμαστε σύντομοι, απλά θα ήθελα να καταγραφεί και η στήριξή μου όπως περιγράφεται και στην έκθεση που εγκρίναμε πέρσι και να πω στον κύριο Σαλαφράνκα, τον φίλο μου, βεβαίως φέτος ο κύριος Φίλε προσπαθεί να βρει μια διαφορετική προσέγγιση λέγοντας πως ε, θα μπορούσε το ζήτημα αυτό να μας απασχολήσει πάρα πολύ στην αρχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αντί για να, είναι, να προηγηθεί της έναρξης των διαπραγματεύσεων και εγώ συμφωνώ με αυτό. Και νομίζω πως έτσι εν μέρη αντιμετωπίζεται και το ζήτημα που αναφέρατε. Βεβαίως, χάρηκα που άκουσα τον κύριο Ποπόσκι και το ότι είναι υπέρ της ε, περαιτέρω ε, ε διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Συμφωνώ και βεβαίω εμείς πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα. και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να θέσουμε αυτό το θέμα και βέβαια οφείλω να συγχαρώ και την κυρία Κοπά που ήταν η συγγήτρια για το θέμα και βέβαια αντιμετώπισε την χώρα σας με βάση κάποιες αρχές λέγοντας πως τα δημιουργή ζητήματα δεν πρέπει να ε, αποτελέσουν εμπόδιο στις ενταξιακές διαδικασίες και όλοι το στηρίξαμε σε αυτό το κοινοβούλιο ήταν μια πραγματικά ε, αντιμετώπιση με βάση κάποιες αρχές και με μακροπρόθεσμο όραμα και θα ήθελα να τονίσω αυτό. Τώρα, να αναφέρω κάποια άλλα ζητήματα. Ο διάλογος ψηλού επίπεδου για την ένταξη νομίζω πως έχει κάποια δυναμική και έχει βεβαίω δημιουργήσει κάποιε προσδοκίε στη χώρα, αλλά είναι κάτι το βραχυπρόθεσμο συμφωνεί ο κύριο Υπουργό Μπορεί να είναι η κατάσταση βεβαίω ε, τώρα διαφορετική σε σχέση με πριν από 12 μήνε, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε αυτόν. Γι' αυτό είναι σημαντική απόφαση τη 10η Δεκεμβρίου. Δεύτερον, να ρωτήσω τον κύριο και αν θυμάται όταν είχε έρθει στα Σκόπια ο Καρλ το υπουργό ε, τότε τη Σουηδία, και είπε τα πράγματα που είπε μόλις ο κύριος Σαλαφράνκα και έκανε τη σύγκριση με άλλες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια όπου υπάρχουν ακόμα συγκρούσεις ή βία και αναρωτήθηκε δημοσίως εάν χρειάζεται να υπάρξει βία πριν αρχίσουν να ασχολούνται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια χώρα. Εγώ ταυτίζομαι με τον Καρλ Μπίλτ και θα ήθελα και ο κύριος Υπουργό να μας απαντήσει, να μας πει πώς αντέδρασε αυτός και οι συναδελφοί του σε αυτή τη δήλωση. Τέλος, σημείωσα στην πρόσφατη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Γκουρεύσκη και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ποπόσκη σήμερα για το ότι είμαστε διεθυμένοι να κάνουμε περισσότερα να υπάρξει κάποιο μνημόνιο συμφωνίας και να έχουμε καλύτερη σχέση με τη Βουλγαρία. Ακούω κάποιους κοινικούς στις Βρυξέλλες που λένε πως ε, τα μέτρα αυτά που προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης ε, από πλευρά Σκοπίων θα φτάσουν μέχρι τον Δεκέμβριο και μετά θα ανακληθούν. Δεν το πιστεύω εγώ, αυτό το λένε κοινικοί, αλλά ο κύριος Γκουρέσκι λέει πως θα συνεχιστεί αυτή η ε, κατεύθυνση της συμφιλίωσης. Και θα ήθελα να το ε, επαναλάβετε και εσείς. Σας ευχαριστώ κυρία Κοπά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Βοβός και πάντοτε ε, είναι ευχάριστο να έρχεστε εδώ να συζητούμε στην Επιτροπή. Τι λέτε για αυτή την ελληνική πρόταση για το μνημόνιο κατανόησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε ικανοποίηση γιατί στην απάντησή σα στην επιστολή αναγνωρίζετε ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη, γειτονικέ σχέσει και να αναβαθμιστούν οι σχέσει συνεργασία με την ε, Ελλάδα. Τώρα, ε, υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Δέχεστε την ελληνική πρόταση. Εάν ναι, πότε θέλετε να ξεκινήσουν, πότε περιμένουν να ξεκινήσουν οι σχετικέ διαπραγματεύσει. Η σε περίπτωση αρνητική, γιατί δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση. Δεν πιστεύετε ότι ε, η σύνταξη και η υπογραφή ενό τέτοιου μνημονίου πρόκειται να συμβάλλει στη δημιουργία ενό θετικού κλίματο, το οποίο πρόκειται να ρωτήσει, ναι, να, αναβοηθήσει στο να επιληθεί το, το πρόβλημα τη ονομασία και πάντοτε όσον αφορά βεβαίω και τι ε, καινούργιε προσπάσει Ευρωπαϊκή Ένωση δια του προσώπου του κυρίου Νίμιτ. Κύριε Κυρίλοφ. Έχω δύο ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι πρόσφατα συναντήθηκα με τον ε, προκάτοχό σας και του υπενθυμίσα πως πριν από 4-5 χρόνια τον είχα ρωτήσει σε αυτή την επιτροπή το γιατί υπάρχει αυτή η δυσανεξία ε, όσον αφορά τους ε, πολίτες τους Μακεδόνες που παίρνουν και βουλγαρική υπηκότητα γιατί υπάρχει μεγάλη ανεκτικότητα για όσους έχουν δεύτερη υπηκότητα κροατική, σερβική, γερμανική κτλ. Και είπε πως αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος. Τον ρώτησα και ρωτάω και εσάς πόσο καιρό περιμένετε να συνεχιστούν αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος γιατί κάποιοι οι οποίοι αισθάνονται ε, πως έχουν βουλγαρικές ρίζες διώκονται και από την επαγγελματική σας δικαιοσύνη. Δεύτερον, πριν από μία εβδομάδα εδώ πέρα είχαμε εδώ πέρα μια διάσκεψη για έναν από τους μεγάλους μας ήρωες, ε, τον Σοτσάροφ, ο οποίος φυλακίστηκε για τις αντιφασιστικές του δραστηριότητες. Αυτό είναι πρόσφατο παρελθόν, όχι μεσαιωνικό και αρχαίο. Ο άνθρωπος είχε γράψει στα βουλγαρικά, είναι γνωστή η ποιησή του. Και μου είπε το γραφείο σας ε, την παραμονή της εκδήλωσης πως αυτό είναι πρόκληση, πως ε, οι Βούλγαροι τον εκτέλεσαν και τώρα τον λένε ήρωα της Βουλγαρίας. Ε, κάτι το οποίο βέβαια είναι αντίθετο με όλες τις δηλώσεις σας πως θέλετε να αναπτυχθεί αυτός ο διάλογος. Αυτές είναι λοιπόν οι ερωτήσεις μου. Ο κύριος ε, Κόβατσεφ, ε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις ε, καλές γειτονικές σχέσεις με την Βουλγαρία. Εμείς σας υποστηρίζαμε πάντα και το μακεδονικό λαό στον δρόμο του προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Αλλά βεβαίως σημασία έχει η ουσία του προβλήματος. Γι' αυτό πρέπει να τα δούμε αυτά. Μέχρι το 1944 οι έννοιες ε, Μακεδονών και Βούλγαρος ήταν ε, συνώνυμες. Τότε έκανε η κομμουνιστική διεθνή στην πρώτη προσπάθεια να χωρίσει τα δύο έθνη και τα κατάφεραν. Ελπίζω η πολιτική των διακρίσεων ε, της, ε, της, ε, της μη ανεκτικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Σκόπια κτλ. να ξεπεραστεί. Είπατε πως ε, δεν έχετε ακούσει οτιδήποτε για διακριτική μεταχείριση Βουλγάρων στη Μακεδονία. Πηγαίνετε και συναντήστε τους ανθρώπους. Φοβούνται να πούνε πως έχουν βουλγαρικά επώνυμα, πως έχουν βουλγαρική καταγωγή. Ο κύριος Μύροσλαβ Ρεζίνσκι παραδείγματος χάρη καταδικάστηκε σε μια τελείως επινοημένη δίκη στη Μακεδονία γιατί είπε πως είναι Μακεδόν Βουλγαρός. Βλέπουμε πως ε, από την κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία του Τίτο και την τωρινή ιδεολογία στα Σκόπια δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και αυτό μας λυπεί. Ε, η Βουλγαρία δεν θα θέσει εμπόδια στην πορεία της Μακεδονίας προς την Ευρώπη, αλλά αυτά τα οποία αναφέρω είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στις Βρυξέλλες, ούτε στη Σόφια. Είπατε ας αφήσουμε την ιστορία στους ιστορικούς, αλλά δεν το κάνετε αυτό. Χρησιμοποιείτε την ιστορία για να φτιάξετε μια εθνική ταυτότητα η οποία είναι προκλητική κατά της Βουλγαρίας. Και ε, ο πρόσωπός σας επίσης είπε κάτι το αρνητικό προσφάτως για ε, τα γειτονικά κράτη της Μακεδονίας που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε με τις δηλώσεις ε, αυτές του εκπροσώπου σας και τι άποψη για την υπογραφή μια συμφωνία σε σχέση με τη δήλωση του 99. Να αδελφοί, άμα συνεχίσετε αυτό το βιολί, δεν θα ακούσουμε απάντηση του Υπουργού. Η κυρία Φαγιόν, Λούνατσεκ, Χρυσόγελος, Νέισκι, γρήγορα γρήγορα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Υπουργέ Ποπόσκη, για την ε, παρουσίαση που κάνατε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ακούσαμε πολλά πράγματα. Ας μην σπαταλάμε το χρόνο μας. Ελπίζω να κρατήσετε όλες σας τις υποσχέσεις σε σχέση με τη Βουλγαρία. Και ελπίζω πως του χρόνου θα υπάρξει και μια επίλυση για το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι ανέφεραν ήδη το θέμα της διαφθοράς. Εγώ θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Τους ετούντες άσυλο που φεύγουν από την Μακεδονία το ερώτημά μου είναι, τι κάνει η κυβέρνησή σας για να περιορίσει αυτό το νέο κύμα ετούντων άσυλο όπως ξέρετε, ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για ένα προσωρινό πάγωμα του καθεστώτος ασύλου ε, και της κατάστασης όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πως τα κάτι μέλη θα μπορούσαν να ζητήσουν ένα προσωρινό πάγωμα για τη Σερβία, τη Μακεδονία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. από όσο ξέρω, δεν είναι μόνο μέλη μειονοτήτων, αλλά και νέοι άνθρωποι που ίσως ποτέ να μην είχαν ε, βρει δουλειά και να πιστεύουν πως θα βρουν δουλειά εδώ. Τι θα κάνετε με τα ταξιδιωτικά πρακτορία που εξακολουθούν να πουλούν εισιτήρια για να βοηθήσουν τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα δυτικά. Πώς εμείς λοιπόν στα δυτικά μπορούμε να δράσουμε ώστε να κάμψουμε αυτό το κύμα μεταναστών που έρχεται από τη χώρα σας, γιατί ορισμένε χώρες δεν είναι ακόμα τμήμα του κοινού συστήματος ασύλου. Ίσως θα μπορούσαμε να περιλάβουμε χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία που είναι ακόμα εκτός, ώστε να εισάγουν αυτό το σύστημα. Έχετε να μας πείτε κάτι για αυτά. Κυρία Λούνατσεκ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε εκ, προ... των Πρασίνων της ομάδας μου κύριε και σε αυτή την συνεδρίαση. Καταρχήν θέλω να πω ότι εξ ονόματος της ομάδας μας είμαστε υπέρ εδώ και χρόνια της έναξης διαπραγματεύσεων της Ένασης με την Μακεδονία και λυπούμεθα πολύ που έχει υπάρξει ε, μπλοκάρισμα από πλευρά της Ελλάδας. Ειλικρινά ελπίζω πως δεν θα γίνει κάτι παρόμοιο από τη Βουλγαρία γιατί το θέμα των διμερών σχέσεων και των προβλημάτων με κράτη-μέλη, ε, κρατη που μπλοκάρουν άλλους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, δεν είναι μέσα στο πνεύμα της Ένωσης. Να αναφερθώ σε δύο θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δέκα χρόνια μετά από τη Συμφωνία της Οχρίδας, οι διεθνικές σχέσεις, διεθνωτικές σχέσεις στη χώρα σας δεν είναι τόσο καλές όσο θα μπορούσαν να είναι υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση και πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε πως αυτό ήδη γίνεται ε, από τα ε, ε, παιδιά, δηλαδή από τις νεαρές ηλικίε. Τι γίνεται λοιπόν στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, από το τοπικό επίπεδο και από την κυβέρνησή σας έτσι ώστε να υπάρχουν ε, μεικτά σχολεία ε, για διεθνωτικά σχολεία. Τι γίνεται με τα σχολικά βιβλία, τα βιβλία ιστορίας, γιατί αν θέλετε να αναπτύξετε μόνο μια καθαρά μακεδονική ταυτότητα για τη χώρα σας, ενώ έχετε τόσες εθνωτικές μειονότητες, είναι κάτι που πρέπει να γίνει αυτό. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τους ομοφιλόφιλους ε, Έχουμε, ε, έχει αποκλειστεί η νομοθεσία σε σχέση με τις λεσβίες και τους ομοφιλόφιλους, ε, τους ε, αμφιφιλόφιλους κτλ. Τι κάνει η κυβέρνησή σας για να καταπολεμήσει αυτή την κατάσταση, όπως έγινε ας πούμε και στην γειτονική σας χώρα, το Μαυροβούνιο, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που ζει στη χώρα σας να ζει χωρίς φόβο. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα είμαι σύντομο. Θέλω να κάνω τρει ερωτήσει. Ο ρόλο κοινωνία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθούσε πολύ και στην ενδυνάμωση τη δημοκρατία και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων και διαφορετικών ομάδων. Έχετε κάποιο σχέδιο για να ενδυναμώσει η κοινωνία των πολιτών που είναι ακόμα αδύναμη στην πρώην κυκλοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Το δεύτερο, το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου μα, αλλά δεν περιλαμβάνεται στα θέματα που συζητάτε στην ενταξιακή διαδικασία και θα έλεγα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μας παρουσιάσετε μια στρατηγική, αν έχετε, για τα θέματα του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον. Και το τρίτο είναι, ε, πράγματι η Ελλάδα στο παρελθόν έχει κάνει πολλά λάθη στο θέμα της ε, προσπάθειας να εξευρεθεί μια κοινή σύνθετη ονομασία. Ε, τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που και η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει μια σύνθετη κοινή ονομασία και νομίζω ότι είναι πιο όριμε και οι δύο κοινωνίε να βρουν μια λύση. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένε πρωτοβουλίε για να το πετύχετε. Νέτσκι. Για, για ένα λεπτό και όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όταν ε, υπεγράφει η δήλωση της ε, χώρας μου πριν από 10 χρόνια ήμουν ε, υπουργό εξωτερικών της χώρας μου και ως κάποια η οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη Μακεδονία θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό εάν έχει ασχοληθεί προσωπικά για τη βελτίωση των σχέσεων με την Βουλγαρία για τα δικαιώματα των υπηκόων εκείνων που έχουν και δεύτερη βουλγαρική ε, υπηκοότητα. Συμφωνώ με την κυρία Λούνατσεκ ε, όταν λέει πως όλες οι βαλκανικές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν λιγότερα προβλήματα αν είχαν περισσότερη συνεργασία. Γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί ορισμένες αρχές και κανόνες και αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Θα, θα προσπαθήσω λοιπόν να τις ομαδοποιήσω, λέει ο Υπουργός, δεν βλέπω κάποια λύση με τόσο λίγο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, η τωρινή κατάσταση και προσθέμενη αξία. Εάν πάμε προς ενταξιακές διαπραγματεύσει και αν δεν πάμε προς τα εκεί. Νομίζω πως τα περισσότερα ερωτήματα τα οποία τέθησαν, ε, περιβάλλον, κριτήρια, τι μπορούμε να κάνουμε για καλές σχέσεις με τους γείτονες, ε, σχετίζονται με το ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρώπη για να ε, εξελιχθούν αυτά τα πράγματα θετικά έχει αποδειχθεί σε όλες τις προηγούμενες διευρύνσεις και το γεγονός πως υπήρχε η ενταξιακή διαδικασία και ότι έπρεπε να ικανοποιηθούν τα κράτη-μέλη με όλα τα κεφάλαια αυτά σημαίνει πως διαμορφώθηκε ε, η υποψήφια χώρα για να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά κριτήρια. Αυτό σχετίζεται βέβαια και με το ερώτημα που αφορούσε το, το περιβάλλον. Έχουμε μια κατάσταση όπου το μέσο το οποίο έχουμε τώρα λέγεται Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. Η Μακεδονία ήταν η πρώτη χώρα η οποία υπέγραψε πριν από 11 12 χρόνια. εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν υποεπιτροπές και η κάθε μία ασχολείται με διαφορετικό θέμα. Π.χ. κράτος δικαίου και δικαιοσύνη, περιβάλλον, οικονομία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου οι περισσότερε από αυτέ τι υποεπιτροπέ δεν έχουν πλέον τίποτα να συζητήσουν γιατί από πλευρά νομοθεσία με το να είμαστε υποψήφια χώρα αλλά να μην έχουμε ξεκινήσει, δεν έχουν τίποτα να μας παρουσιάσουν οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή κοιτάμε το τι εφαρμόζεται στα κρατη Οπότε αν δεν ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις αναρωτιούνται τι θα κάνουν στην επόμενη συνεδρίαση. Και έτσι απαντάμε και στο ερώτημα του κυρίου Χάουιτ για τη βιωσιμότητα αυτής της κατάστασης. Θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων έχει δοκιμαστεί και αφορά κυρίως την ε, διαχείριση κρίσεων. Έχουμε μια κρίση και μετά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε κτλ. Αυτό το οποίο προτείνω στο πλαίσιο της διεύθυνσης και το οποίο θεωρούμε πως χρειαζόμαστε είναι στρατηγική σκέψη και να προλάβουμε τις τάσεις. Ναι, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο των δεξιαγών διαπραγματεύσεων. αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει από πλευρά αποτελεσμάτων με το δικό μας το καθεστώς, δηλαδή 7 χρόνια υποψήφια χώρα, 4 χρόνια ε, συστάσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ε, είναι σχεδόν θαύμα. Κανείς δεν έχει ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση για τόσο πολύ καιρό και να μην ακολουθεί λογική πορεία. Δηλαδή υποψήφια χώρα, μετά ξεκινάνε διαπραγματεύσεις και μετά ε, προχωράμε. Δηλαδή αστευόμενοι μου λένε κάποιοι πως είμαστε τόσο καλή υποψήφια χώρα που δεν θέλουν να μα χάσουν από υποψήφια χώρα. Ε, αυτό είναι εμπόδιο. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση, δηλαδή να έχουμε περισσότερο περιθώριο για τις πιο δύσκολες ε, μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Δεύτερον, διεθνωτικές σχέσεις, η σημασία τους στο περιφερειακό πλαίσιο. Εγώ αυτά θα τα έβαζα μαζί με τα ερωτήματα που έχετε θέσει, π.χ. Ε, άτομα που έχουν βουλγαρική και μακεδονική υπηκότητα ταυτόχρονα. Θεωρώ πως ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο είναι ένας ευρωπαϊκός τρόπος, ε, ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χώρο. Εσείς λαμβάνετε τις αποφάσεις για... Ε, δηλαδή, ο καθένας λαμβάνει τις αποφάσεις για το διαλέγει ποια υπηκότητα θα έχει και το κράτος βεβαίως μετά αναλόγω παρέχει και παίρνει τι αποφάσει. Και αν λάβουμε αυτά τα κριτήρια, προφανώς η πιθανώ η δική μα κατάσταση είναι χειρότερη. Γιατί προς τα εκεί θέμε να πάμε. Εάν ε, ήμασταν όλοι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω πως ε, η μεταχείριση όλων των πολιτών θα ε, ήταν με βάση ευρωπαϊκές αρχές και δεν θα ετίθετο ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης. Θεωρώ πως πρέπει να ισχύσει το κράτος δικαίου κάθε υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με βάση την ουσία της και δεν νομίζω πως πρέπει να μπερδεύουμε τη διαφορά ε, τη συνοριακή εγκληματικότητα και μετά την εθνικότητα, ε, η υπηκότητα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Μεταξύ όσων είναι εντός και εκτός ε, της λέσχης τι θα κάνουμε. Νομίζω πως ήμουν σαφής στο ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε. Πέρα από το ότι έχουμε δοκιμαστεί πάρα πολύ καιρό για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανησυχίες για το ότι η Ελλάδα ανησυχεί για το ότι υπάρχει μια χώρα που λέγεται Δημοκρατής Μακεδονίας ε, στα βορειά της σύνορα και αυτό το χρησιμοποιούν για να μπλοκάρουν τις δεξιακές ε, διαπραγματεύσεις. Θεωρώ πως η μόνη λύση θα ήταν μια λύση που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου. Υπάρχει μια ενδιάμεση συμφωνία του 1995 που ορίζει τους κανόνες επίλυσης του ζητήματος ονομασίας. Νομίζω πως όλοι πρέπει να σεβαστούμε αυτά τα κριτήρια και να τα σεβαστούμε με τρόπο μη επιλεκτικό. Δηλαδή έχουμε ε, το μνημόνιο αυτό συναντήληψης το οποίο οπωσδήποτε βεβαίως ε, έχει κάποιο ε, στοιχείο βεβαίως ε, προκατάληψης και προσπαθούμε να το δούμε με τρόπο που θα είναι μη διχαστικός αλλά πρέπει βεβαίως εδώ πέρα να λάβει υπόψη τις θέσεις και των δύο χωρών και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και να υπογραμμίσω το ότι η Μακεδονία δεν έχει ούτε εδαφικές βλέψεις ούτε θέλει να αλλάξει τα σύνορα ούτε θέλει να αποτελέσει απειλή για κανένα γείτονά τη. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Και η πραγματικότητα νομίζω πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ε, υπογράφουμε συμφωνίες, ε, συντάσσουμε επιστολές ο ένας προς τον άλλον. Τώρα, εάν ε, δεσμευόμαστε για τις υποχρεώσεις μας. Ναι, σαφώς. Είτε μιλάμε για την ενδιάμεση συμφωνία για τη σχέση με την Ελλάδα, είτε μιλάμε για τις ημερείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει στο παρελθόν με τη Βουλγαρία ή με οποιαδήποτε άλλη ε, χώρα ή οντότητα ε, με την οποία έχουμε διμερείς σχέσεις. Αυτά είναι απλώς τα γεγονότα. Και αν τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες νομίζω πως θα ξεπεράσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Πώς είναι δυνατόν να εκκρεμεί αυτό το ζήτημα για τόσα χρόνια. Νομίζω ο κύριος Σαλαφράγκα έφυσε το ερώτημα. Νομίζω πως η ουσία είναι θέμα κινήτρων. Δηλαδή το να είναι κανείς κράτος μέλος ε, είναι πολύ καλή θέση, δεν το αγνοούμε αυτό, έχει δοκιμαστεί νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετά χρόνια. Από πλευρά κινήτρων η θέση μα είναι πω δεν έχουμε υψηλότερη προτεραιότητα από το να λύσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ω εμπόδιο για την ένταξή μα. Οπότε έχουμε σαφέ συμφέρον Και βεβαίω, ε, γιατί όπω είπα, 90% πληθυσμού λέει πω θέλουμε να ενταχθούμε σε αυτά τα δύο κλαμπ. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη θέση, όπως είπαμε, ε, ενός κράτους μέλους που ήδη έχει καταφέρει να παρακάμψει τη διαδικασία λήψη απόφασης για την ένταξη, την έναρξη της συνταξιακής διαδικασίας, ανεξαρτήτως του αν αυτό σέβεται ή όχι αναληφθήσεις ε, υποχρεώσει, αλλά αυτό είναι η άνεση η οποία σας είπα έχει ένα κράτος μέλος. Εγώ θα έλεγα, τηρώντας τη λογική της διαδικασίας διεύρυνση όπως έχει οριστεί εξ αρχής και εστιάζοντας το κοινό μας συμφέρον που είναι να μπουν όλοι στην Ένωση, ε, νομίζω πως θα αυξηθεί η πιθανότητα να ε, βρεθεί μια λύση για το ζήτημα του ονόματος που εκκρεμεί. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε. Δεν θέλουμε εμείς τον εύκολο δρόμο. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία. Σημαίνει 35 κεφάλαια, να ανοίξουν, να κλείσουν συγκρίσεις κτλ. Το κάθε κράτος μέλος, εσείς ως κοινοβούλιο, μπορεί να μας κάνει τη ζωή δύσκολη, εάν δεν εκπληρώνουμε τα κριτήρια, οπότε τα, τα μέσα θα ε, είναι πάντα προς την πλευρά των κρατών μελών, αλλά θέλουμε μια δίκαιη ε, ευκαιρία να μας δώσουν εμάς εξολογήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Το σχόλιο για τον Καρλ Μπίλτ, συγκρούσεις λοιπά Νομίζω πως ε, σε αυτές τις διαδικασίες είναι δύσκολο να τα εξηγήσουμε στους πολίτες, αλλά είναι εύκολο να τα αντιληφθούμε από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό το οποίο είναι ευκολότερο είναι να μην κάνουμε τίποτα και να αγνοήσουμε το ότι ε, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει τα κριτήρια. Αλλά δεν είναι αυτό το σωστό. Νομίζω πως φέτος από όταν γίναμε ε, υποψήφια χώρα έχουμε τις ε, περισσότερες ε, πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα για να απαντήσω και στους κυρίους Κυρίλοφ, Κόβατσεφ, Νέισκι και τη δίωξη Βουλγάρων, ε, τον ε, Μπαπτσάροφ, ε, Τίτο κτλ. Δεν είμαι ιστορικός, ειλικρινά έτσι. Δεν θέλω να αρχίσω να ασχολούμαι την ιστορία εκτός ιστορικού πλαισίου. Γι' αυτό έχουμε προτείνει μια πολύ θετική προσέγγιση, δηλαδή η ιστορία να φεύθει στους ιστορικούς και να φροντίσουμε να μην έχουμε ανάμιξη αυτών των ζητημάτων με την διαδικασία ένταξης. Δεν θα βρεθούν δύο χώρες στη Βουλγαρία, στη, με στα Βαλκάνια που θα συμφωνήσουν σε όλες τις τυχές της ιστορίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να διακινδυνεύσουμε για το μέλλον. Στη δημοκρατία το κράτος δικαίου και ο αλληλοσεβασμός Νομίζω πως πρέπει να πριτανεύσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να μπλοκάρουμε την ένταξη κάποιο τελευταίο. Ε, θέλουμε, μόλις μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποφεληθούμε όλοι. Δεν θέλω να ε, το αναφέρω, αλλά είναι αναπόφευκτο ή, να δούμε πως η διαδικασία ένταξης έχει παρεκτραπεί ορισμένες φορές ε, για να αντλήσουν κάποια ωφέλη σε άλλες τομείς. Και δεν νομίζω πως τα εμπόδια στη δικασία ένταξης θα πρέπει να μπερδεύεται με άλλα ζητήματα τα οποία είναι άσχετα. Και τέλος, η Ευρώπη αφορά τους ε, κανόνες και βασίζεται σε κανόνες και γι' αυτό είναι τόσο επιτυχής. Αν συνεχιστεί αυτό έχουμε μια εγγύηση ε, επιτυχίας. Αλλιώς νομίζω πως διακυβεύεται ολόκληρο το